Euh, chers collègues, bonjour. Excusez-moi de mon retard, mais comme certains d'entre vous aussi. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σας ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά έκανα λάθος στην αίθουσα. Καταρχάς, ας δούμε την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να σας πω ότι μετά τον τρίλογο που είχαμε με το Συμβούλιο για την έκθεση του κυρίου Καστέρ για την ε, ε, Ευρωπαϊκή ε, Χρονιά για την ενεργή, η δραστήρια μάλλον γύρανση που θα είναι το 2012. Είπαμε ότι καταλήξαμε σε συμφωνία 25 Μαΐου κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε, μπορούμε να το βάλουμε μετά το σημείο 19, σαν 19α. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχουν ε, δυσκολίες, άρα το αποφασίστηκε. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση του κυρίου Ρόζα, για το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών, των κοινοφελών ε, κοινωνικών υπηρεσιών μετά την ε, συζήτηση που είχαμε ανάμεσα στους εισηγητέ, στον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητή, εισηγητές αναβλήθηκε η ψηφοφορία μάλλον προτείνεται να αναβληθεί η ψηφοφορία και λόγω του ρυθμού των εργασιών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παράλληλα με τις πρωτοβουλίες του Επιτρόπου κυρίου Μπαγνιέ μέσα στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υιοθετηθεί η έκθεση αυτή στην Ολομέλεια γρήγορα δηλαδή πριν το καλοκαίρι. Επομένως σας προτείνω και όπως ε, σας είπαμε και στο mail ε, στο mail που σας έστειλαν οι συντονιστές προτείνω να έχουμε μια έκτακτη ε, συνάντηση στο Στρασβούργο στις 6 Ιουνίου για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις φαντάζομαι, επομένως ε, και αυτό επιβεβαιώνεται. Τρίτον, τρίτο σημείο, η συζήτηση για το σχέδιο γνωμοδότησης για την, για την πρόκληση που αποτελούν οι offshore πετρελαϊκές δραστηριότητες η δραστηριότητα την εξόριξη φυσικού αερίου, το offshore φαντάζομαι ότι σημαίνει θαλάσσια εξόριξη. Θα το συζητήσουμε σήμερα μετά το σημείο 9 εκεί που λέει για την εμπορική, το σημείο ε, που αφορά την εμπορική η ανισορροπία Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Λοιπόν, με αυτές τις αλλαγέ μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη. Ωραία. Περνάμε στο σημείο 2 και θα ήθελα να σα κάνω πέντε ανακοινώσει την προ... Τι θα θυμόσαστε καταρχάς ότι ε, μας μεταδίδουν, είμαστε web, σε web stream. Επίσης, μέσα στα πλαίσια της κινητοποίησης ε, του Ταμείου Προσαρμογής έπρεπε σε επίπεδο συντονιστών να επικυρώσουμε μια επιστολή που εστάλει στον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμού για τη χρησιμοποίηση του Ταμείου στην περίπτωση της General Motors στο Βέλγιο. Δηλαδή τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να πήραν ένα αντίγραφο της επιστολής αυτής γιατί η Επιτροπή Προϋπολογισμών πρέπει να... Μάλλον όχι πρέπει, ψήφισε ήδη. Α, όχι, λάθος. Ψηφίζει σήμερα για την ε, χρησιμοποίηση του Ταμείου. Ε, ε, τρίτη ανακοίνωση. Στο φάκελό σας θα βρείτε τα πρακτικά των εργασιών της Επιτροπής όταν πήγαμε υπό τη μορφή αντιπροσωπείας στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Θα ήθελα να το διαβάσετε, να διαβάσετε την έκθεση αυτή, διότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η επίσκεψη αυτή για τις εργασίες Επιτροπής μας. Επίσης στο φάκελο θα δείτε και τα πρακτικά με την ανταλλαγή που είχαμε με τον κύριο Λόρι Πέτ που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας για τις εργασίες του στο 2011. Επίσης τα πρακτικά της επίσκεψής μας στην Βαρσοβία. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω και ένα σημείο εξ ονόματος της Επιτροπής μας μαζί με τον κύριο Ρόζας πήγαμε στο Δουβλίνο την προηγούμενη εβδομάδα μέσα στα πλαίσια των τακτικών ανταλλαγών που έχουμε με τις διάφορες υπηρεσίες. Στο Δουβλίνο είναι η υπηρεσία Eurofond και είχαμε πολύ ε, χρήσιμες και πολύτιμες ε, θα τις χαρακτήριζα ανταλλαγές απόψεων και όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας αλλά και για τους μετανάστες. Τους θέσαμε κάποια ερωτήματα που αφορούν την, ε, τις συνθήκες εργασίας τώρα μέσα στα πλαίσια της κρίσης που περνάμε και μας απήντησαν ότι το European War Council, τα εταιρικά συμβούλια, είναι, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξαναδούμε, διότι μέσα στα πλαίσια της κρίσης ε, ε, της οικονομικής κρίσης που περνάμε η χρησιμοποίηση των συμβουλίων αυτών δεν ήταν επαρκής και ο ρόλος τους δεν ήταν επαρκής. Επίσης συζητήσαμε για την κατανομή των, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και είδαμε ότι στην μέση περίοδο ηλικίας, δηλαδή από τα 30 στα 40, η κατάσταση δεν είναι πάρα πολύ καλή. Αυτοί επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Ε, και μα επιβεβαίωσαν και μια αίσθηση που είχαμε ήδη ότι οι πιο ευάλωτοι, αν θέλετε, εργαζόμενοι είναι αυτοί που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση και οι πρώτοι κιόλα. Επίσης, τους ρωτήσαμε για μια πιθανή παρέμβασή τους στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μας είπαν ότι θέλουν να δραστηριοποιηθούν κυρίως στον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί το εξάμεινο αυτό στα κράτη. Ποιες συνέπειες θα έχει σχετικά με τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω τα πρακτικά ούτως ή άλλως υπάρχουν, είναι πολύ πιο λεπτομερή, αλλά έτσι απλώς ήθελα θερμό να σας ενημερώσω για τα τεκτενόμενα. Ε, πάμε στο σημείο 3. Α, πριν φτάσουμε αυτό, θα ήθελετε να προσθέσετε κάτι κύριε Ρόζες για την ε, κατάσταση. Α, όχι. Ε. Με δύο λόγια, οι παρουσιάσεις ήταν πραγματικά πολύ καλές. Όλοι η επίσκεψη ήταν πολύ παραγωγική και όσον αφορά το υλικό αλλά και όσον αφορά τη συζήτηση που έγινε. Κυρίως με εντυπωσίασε η παρουσίαση για το ε, πρόγραμμα CLIP που έχει ε, ολοκληρωθεί και αφορά τη μετανάστευση. Ίσως ε, σε αυτό το τομέα να επανέλθουμε κάποια στιγμή ως Επιτροπή. ίσως ε, ε, και κυκλοφορήσει κάποια, κάποιο υλικό για του, τα μέλη για να θυμηθούν λίγο το θέμα γιατί πραγματικά εκεί γίνονται, ε, διατυπώνονται νέες και καινοτόμες σκέψεις. Ναι, σωστό και αυτό. Πάμε στο σημείο 3. Σας προτείνω να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 13ης και 14ης Απριλίου. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν παρατηρήσεις εγκρίνονται. επομένω, και περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης στην έκθεση για γνωμοδότηση της συναδέλφου Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ για την πέμπτη έκθεση της Επιτροπής για τη Σύνοχη και τη Στρατηγική για την Πολιτική Συνεχής μετά το 2013. Πριν δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια, θα ήθελα να σας προειδοποιήσω ότι για την ε, έκθεση επί της ουσίας στην ε, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουμε ζητήσει να υπάρχει μία παράγραφος για το Ταμείο Προσαρμογής γιατί εκεί δημιουργείται ένα ουσιαστικό πρόβλημα, γιατί διαβάζοντας τον κανονισμό της συνέλευσης, όντως υπάρχει μια οριζόντια αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για να ασχολείται με, το, με τα διαφορετικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής όμως, όμως δεν άκουσα πουθενά, δεν ε, εξακρίβωσε πουθενά ότι το Ταμείο Προσαρμογής για την Παγκοσμιοποίηση εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία ταμείων. Επομένως ε, θα δούμε με την εισηγήτρια πώς μπορούμε να παρέμβουμε, γιατί όντως υπάρχει μια δυσκολία εκεί. Τέλος πάντων, σας δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσετε και τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν στη δική σας έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες, ε, όλους τους συναδέλφους για την συνεργασία τους, ε, κυρίως ε, τους σκιώδεις εισηγητές. 89 τροπολογίες υποβλήθηκαν, πολλές από αυτές εντάχθηκαν σε συμβιβαστικές τροπολογίες. Έχουμε 8 συμβιβαστικές τροπολογίες και υπάρχει και μια καινούργια παράγραφος Πιστεύουμε ότι μπορέσαμε να ε, λάβουμε υπόψη μας ε, το σύνολο των τροπολογιών που υποβλήθηκαν, τέλος πάντων σχεδόν ε, το σύνολο. Τέλος και οι υπόλοιπε πέραν των συμβαστικών τροπολογιών μπορούν να αναλυφθούν υπόψη, μπορούν να γίνουν δεκτέ, διότι νομίζουμε ότι ολοκληρώνουν το νόημα του κειμένου. Λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο. Να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου, όλε τι πολιτικέ ομάδε που εργάστηκαν πάρα πολύ και νομίζω ότι το αποτέλεσμα αξίζει τον κόπο. Ευχαριστώ κυρία Κινιακούντς. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική και ουσιαστική συνεργασία που είχαμε. Τελικά, η έκθεση είναι πολύ ισορροπημένη. Έχουμε περιλάβει όλα τα σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη και αφορούν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 ε, κοινωνική πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τις τροπολογίες να, υπάρξει σχέση ανάμεσα στην στρατηγική του 2020 και την στρατηγική συνοχής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Υπάρχει αυτή η ισορροπία. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία η οποία ε, στηρίζεται στην πρόταση της Elizabeth Shooters, η οποία, την οποία υποστηρίζουμε και η οποία υπογραμμίζει, δίνει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην, ενίσχυση ε, και την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Όλοι νομίζω εδώ συμφωνούμε, όλα τα μέλη της Επιτροπής πιστεύω μπορούν να συμφωνήσουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και θα βοηθήσει και την Επιτροπή Σούρα, δηλαδή να ε, βοηθήσει ε, την προπτική, αυτή την προοπτική του Κοινωνικού Ταμείου εν ώψη και της στρατηγικής 2020. Ευχαριστώ. Και όπως είπε η Φερβάνς, πρέπει να επισημάνουμε ε, τη το θέμα αυτό που αφορά το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης και που ε, αναφέρθηκε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Χίρς. κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους ε, του σκιώδους του Άρντε των Φιλελευθέρων, θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την συγγήτρια για την καλή συνεργασία και είμαστε ικανοποιημένοι από τις συμβαστικές τροπολογίες. Για την τρίτη συμβαστική τροπολογία σχετικά με τις ευάλωτες και μειονεκτικές ομάδες ε, είναι η τροπολογία που τώρα έχει συμπτυχθεί με την τροπολογία ε για τη στρατηγική μετά το 2030. Η στρατηγική τη συνοχή είναι πολύ σημαντική για την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον και για την ανταγωνιστικότητα για να επιτευχθούν οι στόχοι ε, του 2020. Η γνωμοδότηση περιλαμβάνει σημαντικά μηνύματα για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των ε, ταμείων, μεγαλύτερη ορατότητα και για την καλύτερη κατανομή των πόρων στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, λιγότερα διοικητικά άχθη και υψηλότερη διαφάνεια. Θεωρώ ότι ήταν ε, πολύ επικοδομητικό ο διάλογο με την εισηγήτρια και τι άλλε ομάδε και θα ψηφίσουμε υπέρ τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή απασχόληση Ευχαριστώ. κύριε Σχότερ, κυρία Τσίμερ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να επιβεβαιώσω αυτό το οποίο μόλις είπε η συνάδελφος, ότι είχαμε πολύ καλή συζήτηση, πολύ καλές διαπραγματεύσεις. Η συγγήτρια ήταν πολύ ανοιχτή και καταφέραμε να βρούμε τελικά μια πολύ καλή λύση. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για τη συνεργασία. Ευχαριστώ και για την αποδοχή της προφορικής τροπολογίας. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε αυτά που βρίσκονται στη βάση αυτή της έκθεσης και χαίρομαι γιατί καταλήξαμε σε μια κοινή διατύπωση την οποία μπορούν να δεχθούν όλοι. Κατά τα άλλα, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι θα υποστηρίξουμε εμείς ε, τις συμβαστικές τροπολογίες και πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Και η κυρία Τσίμα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Λόπε Φοντάνια για τη δουλειά σας όσον αφορά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για την πέμπτη έκθεση συνοχής. Ήδη αναφέρατε πόσο σημαντικό είναι όλες οι πολιτικές ομάδες να συμμετέχουν και να είναι κοινέ οι τροπολογίες. Αυτό το καταφέραμε νομίζω σε μεγάλο βαθμό και η δική μας πολιτική ομάδα με τις τροπολογίες ε, στο ε, Β, στο Ε και στο ε, H είμαστε ικανοποιημένοι. Ήταν σημαντικές αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που καταβάλλατε για να τις επιτύχουμε. Ως πολιτική ομάδα αποσύραμε τη συμμετοχή μας στην πρώτη συμβαστική λύση γιατί αυτό δεν ανταποκρινόταν στις δικές μας απόψεις Θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να υπάρξει ως μια εδρεωμένη πολιτική και όχι απλώς ως ένα εργαλείο εφαρμογής της στρατηγικής του 2020. Αυτό ήταν το βασικό μας πρόβλημα, το πώς θα εξετάσουμε ε, το θέμα της στρατηγικής για τη συνοχή. Υπήρχαν διάφορες απόψεις στο πλαίσιο της Επιτροπής όσον αφορά την έκθεση αυτή και η αυτονομία του Ταμείου Συνοχής για μας είναι πολύ σημαντική. Θέλαμε λοιπόν η γνωμοδότηση να το αντικατοπτρίζει αυτό και είχαμε την εντύπωση ότι τίθεντο κάποιοι όροι για την πολιτική συνοχής. Μας δόθηκε η εντύπωση ότι θα εξαρτώνται οι πληρωμές από την εφαρμογή, την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής 2020 Μπορεί η τροπολογία 89 να, να απορριφθεί, αλλά θα δούμε τι θα γίνει με την ψηφοφορία για να δούμε μπορεί να ψηφίσουμε αποχή στη συγκεκριμένη τροπολογία. Άκουσα και την προηγούμενη ομιλήτρια, την κυρία Σχόιτε, και υπάρχει και το θέμα του ύψους της συνδρομής στο πλαίσιο των διαθετικών ταμείων. Θα ήθελα να καταλάβω λίγο καλύτερα τι ακριβώς εννοεί η διατύπωση το απαραίτητο ύψος των πιστώσεων. Ο κύριος Ντερόσα και ο Τόμας Μάν. Ένα σύντομο σχόλιο για την παγκοσμιοποίηση ε, και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Νομίζω ότι αυτή η Επιτροπή η δική μας δηλαδή, αλλά και το Κοινοβούλιο εν γέννη. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικό για τον τρόπο που, που θα μπορούσε να να παρέμβει στην λειτουργία του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση. Βέβαια, εντάξει, δεν λέω ότι δεν μπορούμε να το βελτιώσουμε, όμως μην ξεχνάμε ότι η, Ευρώπη θεωρείται αυτή τη στιγμή υπεύθυνη για την κρίση, για την ανεργία, πάντων για όλα τα βάσανα τα οποία περνάνε οι εργαζόμενοι. Το Ταμείο χρηματοδοτεί τα άτομα ε, τα οποία έχουν χάσει τη δουλειά τους. Άρα είναι η μόνη άμεση ε, ε, ενίσχυση που μπορεί να δώσει η Ευρώπη στα άτομα αυτά τα οποία έχουν χάσει την, την δουλειά τους. Επομένω, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνουμε σε αυτό, σε αυτό το Ταμείο Κρίσης γιατί πραγματικά είναι η μόνη βοήθεια που δίνει η Ευρώπη στους άνεργους. Η άμεση δηλαδή, απτή. Ο κύριος Τόμας Μάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τη Βερόνικα για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Όταν έχουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουν όλες οι πολιτικές ομάδες, ε, όταν μπορούμε να βασιστούμε οι μεν δε, ε, βλέπουμε ότι μπορεί να προκύψει ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Υπάρχει μια πολύ σταθερή βάση πάνω στην οποία μπόρεσαν να δουλέψουν οι ομάδες. Ε, και αν δούμε τις διαφορές που υπήρχαν αρχικά, ε, κυρία Τσίμερ, και αν δούμε το τελικό αποτέλεσμα, πιστεύω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο να υπερψηφίσουμε αυτή την έκθεση η στρατηγική του 2020 δεν θέλαμε να αναφέρεται σαν μια στρατηγική απομονωμένη και κάτι το οποίο είναι αόριστο. Θέλαμε να δείξουμε ότι έχει άμεση σχέση με αυτά τα οποία κάνουμε και νομίζω ότι το καταφέρουμε να το δείχνουμε. Και όταν έχουμε επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία είναι υλοποιήσιμα, αυτό το οποίο θέλουμε να δείξουμε είναι ότι θέλουμε απλούστευση, θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς που θέλουν ε, να προωθήσουν έργα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κοινωνικού Ταμείου και των άλλων ταμείων. Επίσης είχαμε προτείνει να έχουμε και κάποιους ε, δείκτες ε, και αυτό έχει γίνει αποδεκτό στις συμβαστικές τροπολογίες ε, και πιστεύω ότι ήταν πολύ θετική εργασία και οφείλεται και στη δουλειά της εισηγήτριας και στη συνεργασία όλων των συναδέλφων. Νομίζω ότι πρέπει να συγχαρούμε όλους για τη δουλειά που έχετε καταφέρει μέχρι τώρα. Très bien. Euh, Madame la si vous voulez conclure la discussion. Ευχαριστώ πολύ. Την εισηγήτρια θα ήθελε να ολοκληρώσει την ε, συζήτηση. Πρόεδρε, προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη μας το νόημα, αν μη τι άλλο, των τροπολογιών. Κάτι το οποίο δεν είναι πάντοτε και εύκολο. Και για την ε, τροπολογία της κυρίας Τσίμερ προσπαθήσαμε να την εντάξουμε στο κείμενο. Χωρίς ε, να αλλάξουμε δηλαδή το νόημα της τροπολογίες της. Κοιτάξτε, δεν θέλουμε να αγγίξουμε τις συμβιβαστικέ τροπολογίες, δεν θέλουμε να αγγίξουμε το συμβιβασμό, δεν, πρέπει να, δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυνο τη συμβαστική αυτή, τη συμφωνία. Επομένως, ε, ό,τι μπορούμε κάναμε και δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία. Ευχαριστώ, κυρία Κομπανιέ. Θα ψηφίσουμε σε λίγο για, την, ε, για τις συμβαστικές τροπολογίες αλλά όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ε, ετοιμάζεται να ψηφίσει η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης την Πέμπτη για θέματα που μας αφορούν. Είδα και τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και την συνθήκη έτσι όπως έχει τροποποιηθεί από την πρόσφατη συνθήκη της Λισαβόνας. Δηλαδή για την δημιουργία του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση όταν αναφέρονται ε, τα διαρθρωτικά ταμεία, το ταμείο αυτό εδώ για την προσαρμογή στην κρίση, στην παγκοσμιοποίηση, συγγνώμη, δεν αναφέρεται. Άρα πιστεύω θα πρέπει να επιμείνουμε στο συνάδελφο να αποσύρει την τροπολογία του, διότι δεν υπάρχει καθήλυν αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για τα θέματα αυτά. Εντάξει, θα πρέπει κάπως ε, ε, να μην προχωρήσουμε σε μια άμεση σύγκρουση, όμως από την άλλη πλευρά είναι και πολιτικό το θέμα. Ε, δηλαδή, εάν παραμείνει αυτή η τροπολογία του κ. Πίπερ στο κείμενο, τότε θα θεωρηθεί ότι η Επιτροπή περιφερειακή Ανάπτυξης είναι η καθήλη αρμόδια επιτροπή για να ασχοληθεί με το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Άρα πρέπει να επιμείνουμε, να το πούμε στον κύριο Πίπερα και εγώ από την πλευρά μου θα κινητοποιήσω τον κύριο Αλάν Λαμασού ο οποίος ε, προφανώς είναι υπεύθυνο λόγω προπολογισμού στα θέματα του Ταμείου Προσαρμογής ε, στην Παγκοσμιοποίηση και ο κύριος Αλέιν ε, θα κάνει και εκείνο κάτι, μια και είναι ο, αυτός ο οποίος συντονίζει αν θέλει τις αρμοδιότητες των επιτροπών για το θέμα αυτό. Άρα θα ήθελα Α, αυτό το σημείο θέλετε να πείτε κάτι. Ζήτησα το λόγο κυρία Πρόεδρε, απλώς και μόνο για να πω ότι θα ήθελα αυτό να γίνει με, με έναν τρόπο που να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο προβληματικός. Αν η Βερονίκ καταφέρει να καταλήξει συμφωνία θα είναι εξαιρετικό. Πάντως συμφωνώ μαζί σας με κυρία Πρόεδρε, να μην δημιουργηθεί προηγούμενο που θα μας βλάψει στο μέλλον όσον αφορά την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ επιτροπών. Άρα συμφωνώ μαζί σας. Ε, πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Πριν να περάσω στο επόμενο θέμα, θα ήθελα να πάμε λίγο πίσω γιατί ε, στις ανακοινώσεις ε, ξέχασα την πιο σημαντική. Να χαιρετήσω την Ελίζα Μπετλίντ, τη συνάδελφο, να της ε, ευχηθώ καλή επιστροφή. Ανησυχήσαμε πολύ, ανησυχήσαμε πολύ. Και πραγματικά το μόνο που μπορώ να σου πούμε, να προσέχεις. Πάμε στο επόμενο θέμα έκθεση της συναδέλφου Edit Bauer για την απορρόφηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, τα συναγόμενα διδάγματα για την πολιτική συνοχή της Ένωσης και ε, στην περίπτωση αυτή θα ασχοληθούμε με τις τροπολογίες. Κυρία Μπάουερ, έχετε το λόγο φυσικά στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής είμαστε στη διαδικασία της συνδεδεμένης επιτροπής ως εμείς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την δυνατότητα να αναφερθώ ταυτόχρονα και στις δύο εκθέσεις, γιατί και οι δύο είναι αλληλένδετες. Αυτό είναι σαφές και ε, από τη φύση των τροπολογιών ένα μέρος αφορά με κάποιες εξαιρέσεις το σύνολο των προβλημάτων. Αναφερόμαστε στα εμπόδια, που, που, εμπόδια στην απορρόφηση. Είναι όμως ε, σαφές ότι οι συνάδελφοι ερμήνευσαν ευρύτερα το θέμα και διείσδησαν τροπολογίες οι οποίες αφορούν μάλλον την έκθεση της Βερόνικας και όχι τη δική μου. Παρά τα αυτά θεωρώ ότι η μεγάλη πλειοψηφία των τροπολογιών για τις οποίες θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους πράγματι διευρύνουν την έκθεση, ε, την ε, κάνουν πιο ακριβή σε κάποια σημεία και άρα η μεγάλη πλειοψηφία των τροπολογιών μπορούν ε, με βρίσκουν ε, σύμφωνοι. Όμως, επειδή για κάποιες παραγράφους έφτασαν πολλές τροπολογίες, θα πρέπει να προχωρήσουμε ε, με συμβιβασμούς 6, 7, 8, 18, 19, 26, 27, ίσως και 22 μπορούν να εγκριθούν εν μέρη 30 ή 36, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 58 επίσης μπορούν να γίνουν δεκτές, 61, 62, 63 επίσης και υπάρχουν και τροπολογίες όπου εισάγονται κάποια νέα στοιχεία όχι όμως κατά ανάγκη στις παραγράφους που αναφέρονται οι συνάδελφοι. Θα προσεγγίσω τους ε, συναδέλφους όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν για να βρούμε μια λύση. Υπάρχουν τροπολογίες που προέρχονται από την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο θέματα Υπάρχουν τροπολογίες που αφορούν και τη γνωμοδότηση της Βερονίκ και τη δική μου. Ε, και η Βερονίκ κατάφερε να καταλήξει σε συμβιβασμούς επειδή ακριβώς υπάρχουν πράγματα που μπορούν να πάνε στη μία γνωμοδότηση και όχι στην άλλη. Υπάρχουν θέματα που ξεπερνούν κατά πολύ το πλαίσιο της γνωμοδότησης και που ουσιαστικά δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο κείμενό της. Θα έρθω λοιπόν σχετικά σε επαφή με τους συναδέλφους σας. Θα ήθελε κάποιος το λόγο? Η κυρία Παπαδοπούλου. Yes. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια εκ μέρους της ομάδας S&D. Διαβάσαμε τις 66 τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Προσωπικά έχω επίσης υποβάλει 9 προφορικές. Ε, περιμένουμε να γίνει αυτή η συζήτηση με την κυρία Μπάουερ ώστε να δούμε πώς μπορούν να ενσωματωθούν στόχος είναι να βελτιωθεί ο τρόπος ε, της ε, υλοποίησης του Ταμείου Συνοχής, κυρίως επειδή τώρα μπορεί να έχει αποτέλεσμα και ως ομάδα θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στις μειονεκτούσες περιοχές και στις περιοχές ε, που είναι σε δυσκολία και πρέπει να βρούμε πραγματικά αποτελεσματικούς κανόνες ε, για την ε, παρακολούθηση του Ταμείου στο μέλλον. Η στενότερη συνεργασία μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής θα βοηθήσει αυτές τις ομάδες. Θέλω λοιπόν να κάνω μια κουβέντα για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε αυτές τις τροπολογίες, γραπτές ή προφορικές, ώστε να μπορέσουμε μπορέσουν να ενταχθούν από την εισηγήτρια σε κάποιες άλλες συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Άλλο αίτημα, άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Α, ο κύριος Ντόμας. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Μέχρι τώρα συζητήσαμε το θέμα της Βερόνικα και υπάρχουν αρκετές συγγένειες. Σωστά είπε η Edith Bauer ότι οι δύο εκθέσεις έχουν κάποιες συγγένειες και θα ήθελα να πω ότι δεν κάνουμε μια απλή γνωμοδότηση αλλά έχουμε το άρθρο 50, δηλαδή έχουμε ίσα δικαιώματα ε, με τις άλλες επιτροπές. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το πούμε για να μην υποχωρούμε ως ε, Επιτροπή Απασχόλησης. Πρέπει να δώσουμε και εμείς τη δική μας διάσταση θα πρέπει και οι άλλε επιτροπέ, δηλαδή να καταλάβουν αυτό το οποίο εμείς διατυπώνουμε. Είναι σημαντικό τομέα και δεν θέλουμε ε, να παραχωρήσουμε τις αρμοδιότητές μας. Δεν κάνουμε δηλαδή μια μικρή γνωμοδότηση. Αυτά τα θέματα των ίσων δικαιωμάτων για μα είναι πολύ σημαντικά. Διαφορετικά θα κάναμε γνωμοδοτήσεις μόνο για τους τομείς για του οποίους υπάρχουν μόνο οι ξεκάθαρε αρμοδιότητε. Υπάρχουν ε, πολλοί στόχοι που μας ενδιαφέρουν στα θέματα της περιφερειακής πολιτικής και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Άλλα στα χέρια της Edith Bauer βρίσκεται σε πολύ καλή θέση αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος κανείς θέλει το λόγο. Όλα καλά. Κανείς δεν ζητά το λόγο. Κυρία Μπάουερ λοιπόν και πάλι σε εσά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να προσθέσω σπουδαία πράγματα. Προφανώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι σκοπεύω να έρθω σε επαφή με τους σιώδεις εισηγητές και όσο όταν χρειάζεται με τους συντάκτες των τροπολογιών όσον αφορά τη συνθήκη υπάρχει είμαστε σε εξαιρετική συνεργασία με την επί αρμόδια επιτροπή και με τον συντάκτη της έκθεσης δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα. Ένα πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχει υπάρχουν εμπόδια στη δυνατότητα απορρόφησης των πόρων και το πρόβλημα ε, που μπορεί να προκύψει είναι ότι και στα περιφερειακά ταμεία και υπάρχουν τα ίδια προβλήματα. Άρα θα είναι δύσκολο να βρεθούν τρόποι ή θα πρέπει να επαναληφθεί το κείμενο ως έχει. Αλλά αυτό μπορεί να δημιουργήσει ε, προβλήματα κατανόησης. Βεβαίως θα βρεθούν οι ε, αναγκαίες λύσεις και θα φροντίσουμε το κείμενο που θα εγκριθεί, που θα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή μας, να εγκριθεί ως έχει ή εν πάση περιπτώσει όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Δεν είπατε αν μπορείτε να συμφωνήσετε με τις τροπολογίες κυρίας Παπαδοπούλου, αλλά υποθέτω ότι θα μιλήσετε κατηδίαν. Εντάξει, οπότε όλοι είναι ενήμεροι και είναι ήσυχοι για την, τις συμβιβαστικές τροπολογίες που θα υποβάλλεται στις 15 Ιουνίου. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 16. Νομίζω ότι τελειώσαμε και με αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης, οπότε φτάνουμε στο σημείο 6 που μας ε, φέρνει στη μελέτη της έκθεσης συναδέλφου πρώην Σιεστερόσα για το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος όπου έχουν υποβληθεί 285 τροπολογίες. Έχετε το λόγο. 285 τροπολογίες, 37 παραγράφους I had written nice short paragraphs and they're becoming they're becoming very large. But anyhow, as we know now, the vote will. Όπως γνωρίζουμε, δεν θα γίνει ψηφοφορία αύριο, θα γίνει στις 6 Ιουνίου, Δευτέρα 6 Ιουνίου, τη Δευτέρα δηλαδή της Ολομέλειας. Εφόσον οι συζητήσει μα ε, στεφθούν από επιτυχία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, επόμενη μια-δύο εβδομάδε, θα είναι νομίζω εύκολη η ψηφοφορία. Η συνεργασία μέχρι τώρα ήταν καλή πρέπει να πω. Έχουμε εντοπίσει τα σημεία στα οποία δίστανται οι απόψεις σε μερικά σημεία μπορούμε να συμφωνήσουμε, σε κάποια άλλα είναι πιο δύσκολο. Θέλω να τονίσω ότι η έκθεση αφορά το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών κοινή ωφελία. Δεν ε, αποτελούν απλώ μια σύνοψη του τι αποτελούν οι κοινωνικέ υπηρεσίε κοινή ωφελία ή το πόσο καλέ είναι. Αυτό που θέλουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει μέλλον για τι κοινωνικέ υπηρεσίε κοινή ωφελία. Γι' αυτό θέλω να ζητήσω από όλου του σκιώδει συζητητέ και από όλου του συναδέλφου να θυμούνται ότι ε, αυτή η έκθεση θα πρέπει να έχει κάποιε προτάσει για το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Διαφορετικά δεν έχει νόημα να κάνουμε μια έκθεση χωρί προτάσεις για το μέλλον. Είναι μια συζήτηση που την έχουμε κάνει πολλές φορές για τις κοινωνικές και κοινή ωφελία και από την τελευταία συζήτηση προέκυψε και ένα φόρουμ πολύ θετικό για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος να συντονίζει τα βήματα τα οποία πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών. Γι' αυτό σε αυτή την έκθεση προσπάθησα να τονίσω την Task Force, την ομάδα εργασίας που αποτελείται από διάφορα μέλη για να προωθήσει ακριβώς τις προτάσεις για το μέλλον. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σε αυτό τον τομέα, ε, σε αυτή την περίοδο κρίσης στην οποία βρισκόμαστε, να τονίσουμε το ρόλο των κοινωνικών υπηρεσιών κοινή ωφελία. Ελπίζω μέχρι αύριο το βράδυ να μπορέσω να έχω ετοιμάσει τη δεύτερη εκδοχή των συμβιβαστικών λύσεων. Έχω δώσει ένα σχέδιο συμβιβαστικών λύσεων και ένα σχέδιο πίνακα ψηφοφοριών σε όλους τους σκιώδεις συζητητές και σε όλους όσους έχουν υποβάλει τροπολογίες και από τις διμερείς απόψεις από τις διμερείς συζητήσεις που έχουμε κάνει ε, με όλους ε, θα γίνουν κάποιες επιπλέον τροποποιήσεις στις συμβιβαστικές τροπολογίες και θα προσπαθήσω μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδος με βάση τις συζητήσεις που θα έχω κάνει με όλους τους σκιώδεις συζητητές και συναδέλφους που έχουν υποβάλει τροπολογίες να είναι έτοιμο ε, το κείμενο για την επόμενη Δευτέρα. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να προσθέσω. προσπαθώ όπου είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε μια σωστή συμβιβαστική λύση. Όπου υπάρχουν λογικές συμβιβαστικέ λύσεις τις αναζητούμε. Υπάρχουν κάποια βασικά σημεία η ανησυχία μας για νομικά ζητήματα και για την ασφάλεια δικαίου. Νομίζω ότι τελικά ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη εξετάζει τους κανονισμούς που αφορούν ε, τις κρατικές συμβάσεις, ήδη εξετάζει τους κανονισμούς που αφορούν ε, τις κρατικές ενισχύσεις και ίσως από αυτές τις αναλύσεις της Επιτροπής προκύψουν αλλαγές στους κανονισμούς. Ε, να μην ε, ε, πούμε λοιπόν ότι είμαστε υπέρ ή κατά κάποιων σημείων που αφορούν νομικά προβλήματα. Να βρούμε μια στάση που δεν θα οδηγεί σε προβλήματα για καμία ομάδα, γιατί ακόμη, όπως σας είπα, εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους κανονισμούς και μπορεί να καταλήξει σε τροποποιήσεις. Είναι εδώ και ο Τόμας Μαν ε, και είναι σημαντικό να το συζητήσουμε ότι δεν θέλουμε να έχουμε κάποιο κανονισμό πλαίσιο στο άρθρο 14 και υπάρχει μια τροπολογία των Πρασίνων που λέει ότι ε, καλό είναι να εξετάσουμε το θέμα του κανονισμού πλαισίου. Στην έκθεσή μου θα παρατηρείτε ότι δεν αναφέρομαι σε κανονισμό πλαίσιο ένας κανονισμός πλαίσιο πιστεύω ότι είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε από πολιτικής πλευράς, αλλά δεν είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε μέσα σε αυτή την έκθεση. Εφόσον υπάρχει καλή θέληση, μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινέ απόψει. Η δική μου ομάδα θα ήθελε να αναφέρεται στην έκθεση ένα κανονισμό πλαίσιο. Αλλά όπω σα είπα, προσπαθώ να ακολουθήσω τη μέση οδό. Προσπαθούμε να βρούμε δηλαδή την ε, κατάλληλη διατύπωση για να ξεπεράσουμε αυτό το σημείο διαφωνίας και να εστιάσουμε την προσοχή μας στο τι πρέπει να κάνουμε στην παρούσα κατάσταση για να διασφαλίσουμε ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινή ωφελία θα παρέχονται στα κράτη-μέλη που έχουν και την βασική αρμοδιότητα για αυτά τα θέματα με τρόπο σωστό. Θέλουμε να ε, παρέχονται σωστά, να είναι ευέλικτες, να είναι φιλικές προς τον χρήστη. Οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τον τρόπο παροχής αυτών των υπηρεσιών και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται αυτές οι υπηρεσίε και οι τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης που αναγνωρίζονται τώρα στη συνθήκη τη Λισαβόνας περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να έχουν θα πρέπει να έχουν δικαιώματα τα οποία θα γίνονται σεβαστά και θα αντανακλώνται τα δικαιώματα των τοπικών αρχών σε αυτό τον τομέα. Πιστεύω ότι υπάρχει η βάση για να δώσει το Κοινοβούλιο μια καλή έκθεση και με βάση τα πρακτικά βήματα που το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν χρησιμοποιώντας το συντονιστικό ρόλο της Επιτροπής και χρησιμοποιώντας τη γνώση που έχουν οι βουλευτές του Κοινοβουλίου σε αυτά τα θέματα και χρησιμοποιώντας τη γνώση που έχουν οι εμπλεκόμενοι στα κράτη-μέλη μπορούμε να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση. Αυτή είναι η πρόθεσή μου, να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε μια καλή έκθεση και ξέρω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες θα βοηθήσουν να καταλήξουμε σε μια σωστή έκθεση. Ευχαριστώ. Κυρία Μπάστος και κυρία Λίντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για όσα είπε. Ε, ξεκαθάρισε και πάλι τη θέση του επ' αυτού του πάρα πολύ ευαίσθητου θέματος των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος σκοπός είναι να βρούμε διατυπώσεις ε, που θα καλύπτουν κάποια θέματα, να προωθηθεί το ζήτημα χωρίς ε, να υπάρχει σημαντική διάσταση απόψεων και διαίρεση επ' αυτού. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει σε επίπεδο, ε, να παρέχονται σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Για μας ποια είναι τα σημαντικά σημεία οι κοινωνικές αυτές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος ποιες είναι κατά την άποψή μας. Έχουν μία πολύ σημαντική διάσταση της ασφάλειας την οποία θέλουμε να σεβαστούμε. Γι' αυτό θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει κανονισμός πλαίσιος ο οποίος θα νομοθετεί για τον τρόπο οργάνωσης ε, ε, λειτουργίας και χρηματοδότησης αυτών των υπηρεσιών. Από την άλλη γνωρίζουμε ότι αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, στην παροχή πρόσβασης ε, σε υπηρεσίες καθημερινής επιβίωσης, γιατί πραγματικά αφορούν την καθημερινή επιβίωση των ευάλωτων ομάδων των πολιτών. Γνωρίζουμε ότι κάθε πρόοδο σε αυτό το θέμα των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το γενικό χαρακτήρα της πρόσβασης ε, σε αυτές τις υπηρεσίες. Πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, ισότητα απέναντι σε αυτή την ε, στην πρόσβαση. Αυτά είναι τα βασικά σημεία βάσει των οποίων ε, είχαμε είχαμε κάποιες επαφές με τους συναδέλφους. Προσπαθήσαμε να εξαλείψουμε κάποιες διαφορές ε, που έχουμε με αυτές τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί. Υπάρχουν συμβιβαστικές θέσεις, προσωρινές, αναμενόμενες, επανεξεταζόμενες, αλλά πολύ σημαντικές. έχουν κατατεθεί σε σχέση με αυτό το σχέδιο γνωμοδότης. Έχουμε σε πολλά σημεία ε, διάσταση απόψεων στο ε, Στη, ακόμα και σε συμβιβαστικές προτάσεις. Πρέπει να διευκρινιστούν τα πράγματα. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε και τη σημειολογία, υπάρχει και το θέμα του task force. Ίσως να είναι υπερβολικός ο μηχανισμός αυτός του παρατηρητήριου. Ένα παρατηρητήριο θα μπορούσε να εξασφαλίσει την συνέχεια αυτών των ε, υπηρεσιών χωρίς να είναι κανένας ε, δυσκίνητος μηχανισμός. Εν πάση περιπτώσει οι επαφές είναι εξαιρετικά παραγωγικές. Περιμένουμε το, την τελική διατύπωση των συμβιβαστικών ε, προτάσεων ο συνάδελ... και από εκεί και πέρα θα κάνουμε κάποιες προσαρμογές για να προσεγγίσουμε τις θέσεις μας σε διάφορα σημεία όπου υπάρχει μεγαλύτερη διάσταση απόψεων. Πρέπει να βρούμε ένα κοινό παρανομαστή για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες, οι διαφορές και βεβαίως ε, θα τις αναφέρουμε ή τις έχουμε ήδη αναφέρει συγκεκριμένα στον ε, εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Ντεύλεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρώσα που διευκρινίσατε ότι δεν συμπεριλάβατε την ε, οδηγία στο παρελθόν. Στο παρελθόν πάντοτε ε, ήμασταν αντίθετοι ως ε, ομάδα, ως ΕΛΚ στην οδηγία πλαίσιο. Θέλω να μιλήσω εκ μέρους του σκιώδους εισηγητή, του κυρίου Μανταμές. Υπάρχουν πολλά συγκεκριμένα ερωτήματα σε αυτή την έκθεση. Είναι πολύ λεπτό το θέμα και οι απόψεις των πολιτικών ομάδων μπορεί να είναι ε, ταυτόσιμες. Είναι ε, λεπτό αλλά και τεχνικό το ζήτημα. Έχει ξεκινήσει όμως μια οικοδομητική ε, προσπάθεια με τη βοήθεια του εισηγητή. Ελπίζουμε ότι οι συμβιβασμοί μπορούν να, να καταταγούν σε τρεις ομάδες. Όσοι έχουν κάποιες συμβιβασμοί είναι καλοί. Για κάποιους άλλους όμως θα θέλαμε αναδιατύπωση. Τέλος υπάρχουν οι T U V και X και Z που, είναι, ε, που δεν μπορούμε να τους δεχτούμε ως έχουν. Επειδή υπάρχει περισσότερος χρόνος τώρα, χρόνος πρέπει να φροντίσουμε το κείμενο να είναι αποδεκτό, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε επί των συμβιβασμών με τον εισηγητή και τους άλλους σκιώδεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμας Μάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι παρόλες τις διαφορές που μπορεί να έχουμε, ε, ε, κύριε Ντερόσα, θέλουμε να έχουμε ένα κοινό αποτέλεσμα. Θέλουμε ε, να έχουμε σημεία στα οποία σε όλη την Ευρώπη συμφωνούμε, αλλά ε, όλα αυτά δεν πρέπει αναγκαστικά να μπουν σε μια οδηγία πλαίσιο, σε σημεία που μπορεί να έχουν την αρμοδιότητα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει η αρχή της επικουρικότητας και υπάρχουν τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης που έχουν μεγάλη αρμοδιότητα, την οποία ε, εφαρμόζουν ε, και εμείς θέλουμε να επιτύχουμε το ότι δεν θα υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός. Θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις ούτε ώστε να μην ε, προκύπτουν στρεβλώσεις σε τοπικό επίπεδο. Και δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα κανονισμό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμφωνώ με τα σχόλιά σα ότι θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι, ότι θέλουμε να δώσουμε πολλέ πρακτικέ συμβουλέ και στι τοπικέ αρχέ αυτοδιοίκηση για το πώ μπορούν να τα εφαρμόζουν στην πράξη αυτά τα οποία ε, προβλέπονται. Και όπω είπε και η Ρεγκίνα Μπάστο, ε, ε, προ αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Υπάρχουν ορισμένε συμβαστικέ λύσει με τι οποίε συμφωνούμε. Με κάποιε άλλε θα θέλαμε να τις τροποποιήσουμε για να τις φέρουμε προς την κατεύθυνση που θα μας βρίσκει σύμφωνους. Δεν υπάρχει μία λύση α, β, γ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε τελικά μία κατάσταση στην οποία θα ψηφίσουμε τις συμβαστικέ λύσεις και θα μπορούν τα κράτη-μέλη και οι τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης να αναλαμβάνουν τις ε, ευθύνες τους σε κάθε επίπεδο. Συνεργασία και συντονισμός, αλλά όχι υποχρεωτική εναρμόνιση. Δεν είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες ε, και ο συνάδελφος Ντερόσα ε, πρέπει να κάτσει να τις δει όλες γιατί υπάρχουν πάρα πολλά, ε, πολλές διαφορετικές ευαισθησίες τις οποίες πρέπει μέσα στους συμβιβασμούς που θα κάνουμε να τις αποδεχθούμε. Ελπίζω ότι θα έχουμε λοιπόν μια πολύ καλή συνεργασία και σας εύχομαι καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Λέει η Πρόεδρος, υπάρχουν άλλα σχόλια πριν δώσω και πάλι το λόγο στον εισηγητή. Θα ήθελα να επισημάνω δύο σημεία προς τον εισηγητή, τα οποία γνωρίζει ήδη, νομίζω δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερη δυσκολία. Αλλά ε, από τις υπηρεσίες μας, ε, από τη γραμματεία μου, ε, επέστησαν την προσοχή σε αυτά τα σημεία. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να εκφράζουμε αιτήματα προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Απευθυνόμεθα προς το θεσμικό όργανο. Νομίζω ότι για την παράγραφο 31 της έκθεσής, της, της σας ε, ισχύει αυτή η παρατήρηση. Και για την παράγραφο 30 ένα παρόμοιο σχόλιο έχω. Και όσον αφορά το φόρουμ για τις κοινωνικές υπηρεσίες ε, γενικού συμφέροντος ή κοινή Ε, αναφέρετε ότι θα θέλατε το επόμενο φόρουμ να οργανωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το να δοθεί εντολή σε εμά στην Επιτροπή Απασχόλησης μια τέτοια εντολή δεν μπορούμε όμως να το κάνουμε θα πρέπει να μιλάμε για το κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο που θα οργανώσει αυτό το φόρουμ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα το οργανώσει η Επιτροπή Απασχόλησης συγκεκριμένα. Αυτές είναι κάποιες ε, παρατηρήσεις ε, νομικής φύσεως που μου επέστησαν ε, την προσοχή οι να τις αναφέρω. Όσον αφορά τις συμβιβαστικές τροπολογίες, θα μπορούσατε να μας πείτε πώς θα οργανώσετε στη συνέχεια τη διανομή τους, πώς θα γίνει ο συντονισμός με τη γραμματεία για να προετοιμαστεί η ψηφοφορία. Τώρα φαίνεται ότι έχουμε χρόνο μέχρι τις 6 Ιουνίου, οπότε μπορούν να προετοιμαστούν σωστά οι τροπολογίες. Ο κύριος Ντερόσα. Καταρχήν σας ευχαριστώ όλους για τα πολύ θετικά σχόλια. Νομίζω ότι υπάρχει η βάση για να έχουμε τελικά μια πολύ καλή έκθεση σε αυτό τον τομέα. Για το θέμα της ομάδας εργασίας της Task Force, συγγνώμη που σαν χαλασμένο γραμμόφωνο ξαναγυρνάω στα ίδια και στα ίδια συνέχεια και επαναλαμβάνομαι, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό που θα δημιουργεί ε, το δυναμικό αλλαγής και βελτίωσης αυτών των υπηρεσιών. Ένα παρατηρητήριο είναι ενδιαφέρουσα ιδέα μεν, αλλά το να έχουμε απλώς ένα παρατηρητήριο που θα παρατηρεί αυτά τα οποία συμβαίνουν δεν προσθέτει κάτι, απλώς θα ήταν επικάλυψη αυτών που ήδη κάνει η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας. Αυτή είναι η εντολή της. το να αντικαταστήσουμε το task force με ένα παρατηρητήριο δεν προσθέτει κάτι στην τωρινή αρχιτεκτονική των μέσων που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα στοιχείο δυναμισμού, ακόμη και στο όνομα αυτού το οποίο προτείνουμε να δημιουργηθεί. Και ε, σε τοπικό επίπεδο, οι εμπλεκόμενοι, οι πάροχοι, οι τοπικές αρχές, όλοι αυτοί με τους οποίους μίλησα από πολλές χώρες, θέλουν να δουν ε, κάτι να κινείται σε αυτό το τομέα. Δεν θέλουν να τα αφήσουμε στην τύχη τους τα πράγματα, ούτε θέλουν να το αφήσουμε σε μεμονωμένες πρωτοβουλίες. Θέλουμε να βρούμε ένα τρόπο ώστε να δημιουργείται μία συνένεση για αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Όσον αφορά τώρα τα νομικά ζητήματα, οι νομικές υπηρεσίες ε, μου έχουν ε, ε, δώσει τις σχετικές παρατηρήσεις. Δεν βλέπω να υπάρχει κανένα πρόβλημα προς το παρόν. Για το αν το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να οργανώσει ένα φόρουμ, το έχω βάλει για δύο λόγους. Ε, ένας λόγος είναι διότι ε, άκουσα από πολλές πηγές ότι υπάρχει, ο κίνδυνος να μην οργανωθεί ποτέ ξανά ένα φόρουμ. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να πιέσουμε να οργανωθεί ξανά ένα φόρουμ γιατί έχει σημασία το φόρουμ για αυτούς που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Το πιο πρόσφατο οργανώθηκε από τη Βελγική Προεδρία και αποτέλεσε μια πολύ καλή πλατφόρμα με 15 συστάσεις για πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και θα ήταν κρίμα και γυρνάω πίσω στην ιδέα που έλεγα για το Task Force. Θα ήταν κρίμα αυτέ οι 15 συστάσει να μείνουν εκεί μέχρι το επόμενο φόρουμ χωρί να κάνουμε τίποτα, ώστε στο επόμενο φόρουμ να πούμε τι δεν κάναμε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ίσως ο Στίβεν ε, να μπορέσει να πει κάτι παραπάνω για το επόμενο σημείο. Από ό,τι θυμάμαι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο παρελθόν είχε οργανώσει μία εβδομάδα σχετικά με την απασχόληση και ήταν κάτι που διοργανωνόταν ε, κάθε χρόνο. Άρα νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα. Δηλαδή, η νομική βάση και ο νομικό μηχανισμό υπάρχει για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να το οργανώσει. Δεν ξέρω αν έχουμε του κατάλληλου πόρου, αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Πάντως ε, πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα ήταν καλό να οργανώσει μια τέτοια εκδήλωση. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην το αφήσουμε να σβήσει σαν πρωτοβουλία. Και γι' αυτό έχω βάλει και μια, μια παράγραφο ε, που λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένα φόρουμ. Δεν αρκεί αυτό όμως. Ε, αν δεν αναλάβει η Επιτροπή τη διοργάνωσή του, θα πρέπει το Κοινοβούλιο να αναλάβει τη διοργάνωση. Θα εξετάσω τη διατύπωση της παραγράφου, αλλά πιστεύω ότι η υπενθύμηση για την οργάνωση του φόρουμ είναι σημαντική. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ωραία. Επομένως, κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορούμε να πούμε ότι η συζήτηση θα γίνει Κύριε Μαν, θέλετε να παρέμβετε και πάλι μετά τον εισηγητή. Ναι, ναι, ναι, το ξέρω, λέει ο κύριο Τόμα Μαν συμφωνώ πρόεδρε το θέμα σχετικά με την απασχόληση και την ανεργία δεν ήταν το βασικό θέμα της έκθεσης αλλά μετά από αυτά που είπε ο εισηγητής θα ήθελα να πω και να το συζητήσουμε στους συντονιστές ε, γιατί είχαμε την ε, εβδομάδα για την ανεργία ήταν μια εβδομάδα που διεξήγεται την εβδομάδα του Στρασβούργου την εβδομάδα της ε, Ολομέλειας ήταν αυτή η εβδομάδα της ανεργίας που διοργανώθηκε διοργανωνόταν στι Βρυξέλλες. Και δεν είχαμε καμία δυνατότητα να συμμετάσχουμε γιατί ήμασταν στο Στρασβούργο. Εμεί θέλουμε μια τέτοια εβδομάδα στην οποία να υπάρχουν και ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει και άνεργοι οι οποίοι ίδιοι να λένε ε, πώ έφτασαν στην ενεργεία και πώ από την ενεργία ξαναπέρασαν στην απασχόληση. Ήταν σημαντικό να έχουμε την αυθεντική μαρτυρία των ίδιων των ανθρώπων. Ένα τέτοιο φόρουμ είναι ενδιαφέρον. Είναι κάτι το οποίο παλέψαμε να έχουμε, Στίβεν, και γι' αυτό ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε, που έλαβα το λόγο και πάλι. αυτό το θέμα για την εβδομάδα της ανεργίας ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς είμαστε εκπρόσωποι του λαού, των πολιτών της Ευρώπης και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία γιατί είναι και καθήκον μας να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να πούμε εμεί τίποτα. Αυτού πρέπει να αφήσουμε να μιλήσουν. Εμεί είμαστε απλώ οι υποστηρικτέ του. Και είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον να, να ακούσουμε τη φωνή των πολιτών. Αυτό ήθελα να πω σε μια σύντομη παρέμβαση. Ευχαριστώ δεν έχουμε πάρει καμία αντίρρηση, γιατί ούτως ή άλλως είναι συμπληρωματικό το θέμα και έχουμε και χρόνο. Α, τώρα ξαναρχίσαμε στη συζήτηση, διότι και ο, και ο Steve μου ζητάει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ήθελα να πάρω το λόγο, αλλά μια και ε, συζητάμε την δυνατότητα εμείς να αναλάβουμε δράση σε σχέση με, το, με την ανεργία. Να σας πω ότι για χρόνια ολόκληρα ε, παρεμβαίναμε στην οργάνωση της εβδομάδας ανεργίας. Ε, Ήταν μια ανεξάρτητη οργάνωση, η, οποία το, η υπηρεσία η οποία το οργάνωνε. Τέλος πάντων κάποια στιγμή αποσύραμε την υποστήριξή μας, διότι τελικά οργανώναμε αυτή την εβδομάδα ανεργία στην ε, εβδομάδα του Στρασβούργου. Μια και έχω το λόγο τώρα, θα ήθελα εν συντομία σε σχέση με την πρόταση που έγινε για τη δημιουργία μιας task force για τις δημόσιες υπηρεσίες, να σας πω ότι υπάρχει ένα προηγούμενο. Θα θυμόσαστε ενδεχόμενο, κυρία Πρόεδρε, ότι πριν από μερικά χρόνια είχε γίνει ένα φόρουμ ε, για την εταιρική ευθύνη όπου συμμετείχαν ε, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου και, τις, ε, και εμείς ε, συνεισφέραμε ενεργά. Επομένως νομίζω ότι μπορούμε να το υποστηρίξουμε εκ νέου. Πολύ ωραία, λέει η Πρόεδρος. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό της σημερίσιας διάταξης. Και όπως είπαμε, η συζήτηση για τις τροπολογίες, τις συμβαστικές τροπολογίες και η ψηφοφορία θα λάβουν χώρα στις 6, 6 Ιουνίου μέσα στα πλαίσια μιας έκτακτης συνεδρίασης στο Στρασβούργο. Περνάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Είναι η γνωμοδότηση που σας ζήτησα για την εντολή για τον τριμερή διάλογο σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού 2012. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες διότι οι περισσότερες είναι πάρα πολύ χρήσιμες και επιτρέπουν να καλύψουμε πολλά σημεία σημεία που αναφέρονται στο σχέδιο γνωμοδότησης. Για την τροπολογία της 1 της κυρίας Μαρκίνα, εγώ συμφωνώ απόλυτα, δεν υπάρχει καμία δυσκολία. Για την τροπολογία 2, η οποία υπευλήθη από την κυρία Φιγκερέντο, και τον κύριο Γιαρίκ. Δεν έχω αντίρρηση. Αφορά την ανάγκη να συνεχίσουμε τη μελέτη για τις συνθήκες ε, διαβίωσης των αποσπασμένων εργαζομένων, να δούμε τα μεταναστευτικά ρεύματα. Σε αυτό το θέμα να σας πω ότι υπάρχει ένα σχέδιο πιλότος για την οδηγία από, για τις αποσπάσεις. Ε, υπήρχε μια χρηματοδότηση για το 2010, έγινε μια μελέτη μάλλον το 2010 και τα αποτελέσματα της μελέτης θα τα έχουμε μέχρι το τέλος του έτους. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι οι τροπολογίες που υποβλήθηκαν ε, ζητάνε από την Επιτροπή να μπορεί να συνεχίσει την παρακολούθηση των, της εφαρμογής της οδηγίας και να δούμε πώς ολοκληρώνονται τα μεταναστευτικά ρεύματα. Η τροπολογία 3 της κυρίας Αρκίνα αφορά αυτή την ιδέα ότι λαμβάνοντα υπόψη τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πρέπει κάποιες ενέργειες να λάβουν χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άλλες σε εθνικό επίπεδο και δεν θα πρέπει να είναι αντιφατικές αλλά να οδεύουν προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό είναι το πνεύμα της τροπολογίας νομίζω. Εγώ θα πρότεινα μια συμβιβαστική τροπολογία για να ε, τονίσουμε περαιτέρω την συμπληρωματικότητα των δράσεων και τη συγκρισιμότητα των δράσεων. Διότι υπάρχουν οι δαπάνες ε, που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη για να ε, συνοδεύσουν αν θέλετε μια κάποια δυναμική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται συνέχεια ε, στον τρόπο με τον ε, που υποβάλλονται οι προπολογισμοί. Δεν υπάρχει κάποια συγκρισιμότητα, κάποια δυνατότητα συγκρισιμότητα. Δηλαδή, αν θέλουμε να δούμε ποια είναι τα χρήματα τα οποία δαπανώνται για την εκπαίδευση, εκεί έχουμε δυσκολίε. Γιατί είναι διαφορετική η τυπολογία, αν θέλετε, των προπολογισμών. Αυτό είναι μια προσπάθεια μακροπρόθεσμη. Όμως εγώ έχω ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και θα συνεχίσουμε να, την εργασία μας με την, συνεργασία μας με την κυριαρχή. Τώρα, ε, τροπολογία 4 Κάσλερ. Επαναλαμβάνει τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε μέσα στα πλαίσια του τριλόγου για την ε, δραστήρια η ενεργή γύρανση αν θέλετε και το ευρωπαϊκό έτος ε, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό όπω είχαμε πει και στην αρχή. Η τροπολογία 5 της κυρίας Αρκίν. Εδώ ζητάμε από τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε μια μεγαλύτερη περαιτέρω ε, συνεργασία ε, όμως θα πρέπει κυρία Χάρκιν να τονίσουμε ότι ναι μεν πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία όμως δεν υπάρχει σύμπτωση, πλήρης σύμπτωση. Αυτός ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης θα πρέπει να παραμείνει και αυτό θα εμφανιστεί και στην τροπολογία την οποία θα ψηφίσουμε. Τροπολογία 6 της κυρίας Φιγκερέντο και του κυρίου Γιάρικ για το θέμα του βάρου συγχρηματοδότησης όταν τα κράτη-μέλη δηλαδή αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Είναι μία ιδέα την οποία δεν μπορέσαμε να επικυρώσουμε όταν διορθώσαμε, αν θέλετε, την λειτουργία των διορθωτικών ταμείων ε, μέσα στα πλαίσια της κρίσης. Δεν θέλουμε να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν ε, αργότερα μόνο την, ε, το, το κομμάτι της χρηματοδότησης, αλλά θα πρέπει και το ποσοστό, το ποσό της χρηματοδότησης να είναι μικρότερο. Επομένως εδώ οι συγγραφείς της τροπολογίας αυτής προτείνουν να πούμε ότι η συμμετοχή των κρατών μελών δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 10% της αξίας των 10 project αυτών. Εγώ προτείνω μια προφορική τροπολογία που θα λέει ότι η συμμετοχή των κρατών μελών αυτών δεν θα έπρεπε μάλλον θα, ή θα έπρεπε να περιοριστεί στο 10% της αξίας των project. Δεν νομίζω ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα. Πάμε στην τροπολογία 7 της κυρίας Τούρινεν και εδώ συμφωνώ αναφέρεται στις νέες πηγές ε, εισοδημάτων που θα μπορούσαν ε, να χρηματοδοτήσουν τον κοινωνικό προϋπολογισμό. Άρα με τον τρόπο αυτό θα υπάρξουν και πόροι για την κοινωνική ένταξη κτλ. Τροπολογία 8 του κυρίου Ούρη ε, προτείνει να επαναδιατυπώσουμε τις ε, προϋποθέσεις συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων και να διαδώσουμε τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την μετεκπαίδευση των απολυμένων εργαζομένων κτλ. Εγώ συμφωνώ, απλώς σου λέω να συμπληρώσουμε το κείμενο αυτό. Ε, τονίζοντας τα θέματα αναδιάρθρωσης των εταιριών, των επιχειρήσεων. Συγγνώμη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παραμείνει. Γιατί ο, κύριο Συνάδελφο Ούρη λέει ότι θα πρέπει τα θέματα αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων να μην αναφερθούν. Κάτι το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνη. Η τροπολογία 9 του κυρίου Φιγκερέντο και Γιάρικ ε, προτείνουν να υπάρχει μια συγκεκριμένη δημοσιονομική γραμμή για την ε, μετατροπή της ε, πρόσκαιρης εργασίας σε κάτι πιο μόνιμο. Υπάρχει αυτό το project pilotos στο οποίο αναφερθήκαμε. Θα μπορούσαμε ίσως από την ΚΟΕ να ζητήσουμε να αποσύρει την τροπολογία αυτή. Και θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Τώρα, η τροπολογία 10 του συναδέλφου Τσάμπα Ούρη Υπάρχουν πολλοί φάκελοι τους οποίους δεχόμαστε. Επομένως, την τροπολογία αυτή συγκεκριμένη δεν μπορούμε να την ε, δεχτούμε. Και εφιστώ την προσοχή των συναδέρφων για την τελευταία περίπτωση για το Ταμείο Προσαρμογής για την ε, Παγκοσμιοποίηση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό θα έλεγα ε, οι νέες τεχνολογίες, ε, οι θέσεις ε, πράσινης απασχόλησης. Πιστεύω ότι αυτά είναι μέσα για να βρεθεί ένα, ένας τρόπος να καλύψουμε το έλλειμμα, αν θέλετε, θέσεων απασχόλησης. Έτσι νομίζαμε. Όμως τελικά στη Δανία ήταν, βρέθηκε μια πρόφαση για να ε, καταργηθούν, ε, μεγάλος αριθμός θέσεων απασχόλησης σε μια επιχείρηση η οποία ασχολείται με την αιωλική ενέργεια και η οποία μετακόμισε στην Κίνα. Επομένως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί διότι δεν μπορούμε να καταργούμε κάτι και μετά να ε, μην καλύπτουμε ας πούμε τα κενά που μπορεί να, μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τώρα, η τροπολογία 11 με βρίσκει σύμφωνη. Τούρινεν Κορνέλισεν. Γιατί μας δίνει μια δυνατότητα να, να αντιμετωπίσουμε, να σταματήσουμε τις ε, συλλογικές ε, απολύσεις περιορίζουμε τις απώλειες δηλαδή. Η τροπολογία 12 του Ρίνεν και Σρέτερ είναι μια τροπολογία που ενδυναμώνει την, ε, το κείμενο και τις νομοθετικές διατάξεις ε, και ε, που αφορούν και το πρόγραμμα Progress όσον αφορά το, την εφαρμογή της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού, άρα το, δεχτώ, το μπορώ να τη δεχτώ. Τροπολογία 13 Φιγκερέντο, κυρίας Φιγκερέντο και ε, του κυρίου Λεγιαρίκ. Αυτή η τροπολογία μου δημιουργεί ένα κάποιο πρόβλημα, διότι προτείνουν η συμμετοχή των κοινωνικών οργανώσεων, ε, η χρηματοδοτική συμμετοχή των κοινωνικών οργανώσεων σε έργα που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10%. Είναι μια τροπολογία που εντάσσεται στην ίδια, ε, στο ίδιο πνεύμα ε, με την τροπολογία 6 αλλά το, η τροπολογία 6 που αφορούσε το Ευρωπαϊκό Ταμείο, Κοινωνικό Ταμείο δεν μου δημιουργού, τα, γενικά τα κοινωνικά ταμεία στην, ε, στην Ευρώπη δεν με έβρισκε αντίθετη. Εδώ όμως, μια και μιλάμε για το progress, εδώ πιστεύω ότι η τροπολογία αυτή δημιουργεί προβλήματα. Τώρα η τροπολογία 14 των ιδίων ε, συγγραφέων, εδώ εκφράζεται η λύπη για τις πενιχρές πιστώσεις του προπολογισμού για τα επιμέρους τμήματα του προγράμματος Progress. Εδώ δεν έχω αντίρρηση. Τροπολογία 15 των ιδίων συγγραφέων. Εδώ ζητάνε την, ε, τον διπλασιασμό των ε, πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ε, αυτό εντάσσεται στο πνεύμα των συζητήσεων που είχαμε τον Επίτροπο και ίσως θα έπρεπε να εξακριβώσουμε με την εισηγήτρια επί της ουσίας, την κυρία Μωράν Σαρτιέ, για να δούμε πώς μπορεί να ενταχθεί η τροπολογία αυτή στην γνωμοδότηση. Ναι, όντως νομίζω ότι καλό είναι που το εντάσσουμε τώρα, διότι μέσα στα πλαίσια της εντολής για τον τρίλογο αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Αλλά θα πρέπει να το εξακριβώσουμε, να δούμε πώς δηλαδή θα γίνει η διατύπωση, θα πρέπει να συνεργαστούμε με την ε, καθήλυνη εισηγήτρια, αρμόδια εισηγήτρια και μετά θα το επαναδιατυπώσουμε το κείμενο. Τροπολογία 16 δική μου, ε, θέλω να συμπληρωθεί η παράγραφος 8 και να μιλήσουμε για τη δημιουργία μιας κατηγορίας ενδιάμεσων περιοχών. Είναι νέο το θέμα και νομίζω ότι εδώ είναι χρήσιμο η Επιτροπή μας να πει την άποψή της, διότι πολλές ε, περιφέρειες θα ενδιαφερθούν, πιστεύω, με αυτή τη νέα ε, κατηγορία. Τώρα, τροπολογία 17 του κυρίου Όρη προτείνει να διαγραφεί η αναφορά στη μείωση του αριθμού των ατόμων που πλήττονται ή που απειλούνται από την φτώχεια. Εάν ο κύριος Όρη ε, συμφωνεί να το συνδυάσουμε με, τον, ε, με την τροπολογία 18 του κυρίου Γιοβίνα. Θα μπορούσα να δεχτώ τις, ε, την ε, αλλαγή της στην επαναδιατύπωση, αλλά να μην γίνεται, να μην διαγραφεί η αναφορά στην φτώχεια. Ο κύριος Γιοβίνα αναφέρει ποιες είναι αυτές οι ευάλωτες ομάδες. Εγώ προτείνω να διαγραφεί η αναφορά στους Ρωμά, γιατί πιστεύω ότι τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάλλει μια πρόταση για το θέμα αυτό, α, πιστεύω μάλλον λάθος, ότι θα έπρεπε να παραμείνει η, η αναφορά στους Ρωμά. Τώρα, πάμε στην τροπολογία 19, Φιγκερέιντο Λεγιαρίκ. Εδώ αναφέρεται ε, προτείνεται να συμπεριλάβουμε και την διάσταση του φύλου. Αυτή είναι μια τροπολογία πάρα πολύ καλή που μπορούμε να υποστηρίξουμε. Τροπολογία 20 Χαρκίν ε, επαναλαμβάνει την ε, υποστήριξή μας στην χρήση του μηχανισμού της, των μικροχρηματοδοτήσεων. Συμφωνούμε και εδώ. Η τροπολογία 21 του Ρίνεν αναφέρεται στην, στις πράσινες θέσεις απασχόλησης. Εγώ θα έλεγα ίσως να βρούμε ένα συμβιβαστικό κείμενο, γιατί για άλλη μια φορά δεν πιστεύω ότι όλες οι πράσινες θέσεις απασχόλησης είναι ε, σωστές θέσεις, ε, αξιοπρεπείς θέσεις, γιατί ο στόχος μας είναι να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης μέσα στα πλαίσια των πράσινων θέσεων απασχόληση. Τέλο πάντων θα πρέπει να βρούμε έτσι μια πιο μια καλύτερη διατύπωση. Τροπολογία 22 της κυρίας ε, Τούρινεν πάλι, συμφωνώ, με βρίσκει σύμφωνη. Πολύ καλή τροπολογία που αναφέρεται κυρίως στην ανεργία των νέων και που ζητάει μια μια παρέμβαση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Τροπολογία 23 του Τσάμπα Ούρη. Λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί ο κύριος Όρη δεν είναι εδώ. Εγώ θα ήθελα να το συζητήσω μαζί του γιατί ζητάει την διαγραφή αυτής της παραγράφου 10 που αναφέρεται στην ε, ανάγκη να υποστηρίξουμε ε, τους εταίρους μας της περιοχής Μεσογείου στην αναμόρφωση των αγορών εργασίας και του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, μια πραγματική πρόκληση ε, και αυτό το είχαμε πει και όταν πήγαμε να επισκεφθούμε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Είδαμε ότι είναι πολύ μεγάλη συνεισφορά που θα μπορούσε να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει στην ολοκλήρωση στην, και στην ενδυνάμωση του κράτους, του κράτους δικαίου σε αυτή την περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει να τονίσουμε τον, λόγο, τον ρόλο του κοινωνικού διαλόγου, των συλλογικών συμβάσεων και της σωστής οργάνωσης της αγοράς εργασίας. Ελπίζω ο κύριος Όρη θα δεχτεί είτε να επαναδιατυπώσουμε το σημείο 10 ή θα να απορρίψουμε την τροπολογία 23. Τροπολογία 24, δική μου τροπολογία. Θέλουμε και εδώ να Πρόκειται για μια τροπολογία που είναι αντίθετη από την τροπολογία 23, διότι ενισχύει μια διάσταση την οποία νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε για τις ε, χώρες του Νότου, για, τις, μάλλον για, τους, ε, ε, για την περιοχή της Μεσογείου εν γέννη. Η τροπολογία 25 συνδυάζεται με την τροπολογία 24, διότι και εδώ αναπτύσσεται ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση αγοράς εργασίας. Η τροπολογία 26 αφορά μια νέα παράγραφο που σας προτείνω να προσθέσουμε και που αφορά την Ευρωπαϊκή Πολιτική Υπηρεσία. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ζητηθεί επί μακρόν σε, κοινοτικό επίπεδο και τελευταία τροπολογία είναι η τροπολογία 27 του Φιλίππου Μπουλό που αφορά την χρηματοδότηση για την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων και το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Θα θυμίσω ότι είναι εισηγητής για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ο κύριος Μπουλό, επομένως η τροπολογία του μπορεί να είναι χρήσιμη. Όμως θα πρέπει να διευκρινίσουμε αυτή τη στιγμή το τι θέλουμε να χρηματοδοτηθεί διότι το να χρηματοδοτήσουμε έτσι γενικά την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων είναι ένα project πιστεύω ιδιαίτερα φιλόδοξο και δαπανηρό. Αν θέλουμε δηλαδή να παραμείνουμε έτσι τόσο ασαφείς στην διατύπωση. Τώρα από εκεί και πέρα οι συνάδελφοι μπορούν να υποβάλουν και άλλες προτάσεις. Νομίζω ότι υπήρξα ε, πολύ λεπτομερής στην παρουσίαση των τροπολογιών, αλλά μια και έχουμε χρόνο, κατ' εξαίρεση, εποφελήθηκα για να σας παρουσιάσω ε, και ουσιαστικά πλέον τις τροπολογίες και όχι να μην περιοριστώ στο είμαι υπέρ ή κατά κάποιων τροπολογιών. κύριος Τόμας Μάν. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι πολύ σωστά χρησιμοποιήθηκε ο χρόνος και η πρόεδρος της Επιτροπής καμιά φορά μπορεί να πάρει και λίγο περισσότερο χρόνο. Νομίζω ότι ήταν ένα σημαντικό τομέα και αξίζει τον κόπο να κάνω αυτή τη συζήτηση. Όσον αφορά το σημείο 10 είναι σημαντικά αυτό που είπε ο συνάδελφο Τσάμπα Όρη σχετικά με τι πιστώσει ε, πληρωμών. Ε, νομίζω ότι ε, πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώ συμβαίνει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή για την Παγκοσμιοποίηση παραμένει όπως ε, είχε όταν ε, το θέσπισε ο πρόεδρος ε, Μπαρόζο και ποιες είναι οι σχέσεις και με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Νομίζω ότι αυτό το οποίο αναφέρεται ότι πρέπει να δοθούν πόροι με βρίσκει σύμφωνο και αυτό που προτείνει ο κ. Τσαμπαόρη είναι σωστό. θέλουμε ε, να δούμε ποια ονοματολογία χρησιμοποιείται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής για την ε, παγκοσμιοποίηση και πιστεύω ότι αυτή η τροπολογία ε, θα έπρεπε να είναι αποδεκτή. Συμφωνώ και στο σημείο 12 το Ρόνεν και Σρέτερ για το θέμα του Progress το Progress, το κοινωνικό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη, ε, είναι πολύ σημαντικό τομέα και δεν δίνουμε ε, τα κατάλληλα μέσα. Και αν ε, δοθούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ όπω είχε σκεφτεί, και εγώ είμαι στην Επιτροπή Προπολογισμού και θα προσπαθήσουμε να το επαληθεύσουμε, αλλά πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε ένα σημαντικό μήνυμα. Όσον αφορά την τροπολογία 15 για το διπλασιασμό του Ταμείου. Ναι, αν είχαμε χρήματα, καλά θα ήταν να το κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι πολύ αποτελεσματικό, πολύ πιο αποτελεσματικό από πολλές άλλες, αποτελεσματικότερο από πολλές άλλες πρωτοβουλίες. Συμφωνούμε λοιπόν να το υποστηρίξουμε, αλλά τώρα να το διπλασιάσουμε θα πρέπει να δούμε το συνολικό πακέτο. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα μεμονωμένο σημείο στο οποίο θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα. Θα δούμε, πρέπει να δούμε και τις επιπτώσεις για άλλους ε, τομείς. Και δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση από πλευρά κρατών μελών να αυξήσουν τα μέσα που διαθέτουν. Λόγω της κρίσης καταλαβαίνετε ότι τα κράτη-μέλη έχουν πολλές δυσκολίες. Ε, και υποστηρίζω και την τροπολογία 24 την οποία θεωρώ σωστή και ίσως ε, μαζί με την 23 θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε. η δημοκρατική δομή του διαλόγου θα πρέπει να συνεχιστεί και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και με βρίσκει ε, σύμφωνο. Και το 26, η τροπολογία 26 είναι επίσης πολύ σημαντική το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πολιτικής Υπηρεσίας δίνει στους νέους την πρωτοβουλία να κάνουν κάτι και τους δίνει και τα κίνητρα, τους δείχνουν ότι είναι χρήσιμοι, ότι κάποιος τους χρειάζεται και επομένως έχουν λόγο να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν για να συνεισφέρουν. Δεν μπορώ εγώ να μιλήσω στη θέση του Τσάμπα Ορή, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία οι τάσει είναι σωστέ. Αυτά ήθελα να πω και σα είπα ποιε είναι οι τροπολογίε με τι οποίε συμφωνώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε και για την παρατήρησή σας και για το πνεύμα με το οποίο προσεγγίζετε την έκθεση αυτή. Κυρία Τούρνεν. Ευχαριστώ. Εγώ θα μιλήσω δανέζικα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τη σημαντική αυτή γνωμοδότηση που αφορά τον προπολογισμό του 2012. Συνολικά πιστεύω ότι συμφωνούμε. Στόχος είναι να δοθεί ένας προϋπολογισμός που θα στηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, πράσινων θέσεων εργασίας που θα ενισχύουν τον, την κοινωνική ένταξη. Και είμαστε πιστεύω έτοιμοι για, να, γίνει, να επέλθει συμφωνία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η συμφωνία να αφορά και τις τροπολογίες που αν δεν κάνω λάθος είναι 21. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν είναι πολύ ε, συγκεκριμένες. Η 21 δεν είναι πολύ συγκεκριμένη. Η 23 τώρα για τη Βόρεια Αφρική. Συμφωνούμε είναι σημαντικό το θέμα και είναι και θέμα αλληλεγγύης. Δεν συμφωνώ με τον Örη για αυτή την πρόταση διαγραφής. Να μην ξεχνάμε ότι το Μάρτιο η κυρία Άστον συνέταξε ένα σημαντικό πρόγραμμα για τη νέα πολιτική γειτονία και ένα μέρος του αφορούσε την δημιουργία θέσεων εργασίας τη βελτίωση της αγοράς εργασίας. Λοιπόν, ακούγεται περίεργο η Επιτροπή ε, Απασχόλησης να μην στηρίζει αυτή την ιδέα. Τώρα, τελευταία ιδέα. Για μας τους πράσινους είναι σημαντικό να υπάρχει, να είναι ρεαλιστική η πρόταση του προϋπολογισμού. Δεν αφορά τεράστια ποσά, δυστυχώς. Υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί και τώρα πρέπει να παλεύουμε για κάθε ευρώ που επιθυμούμε. το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να διπλασιαστεί. Αυτό είναι όνειρο που δεν είναι ρεαλιστικό. Από πού θα έρθουν τα, τα χρήματα. Πρέπει να μην βάζουμε λοιπόν τόσο φιλόδοξους στόχους. Οι στόχοι μας να είναι ρεαλιστικοί και να είναι και ε, ρεαλιστική η περιγραφή της των πόρων. Πρέπει όμως να στηρίξουμε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μήπως θέλει η Κομισιόν να πάρει το λόγο στο πλαίσιο του προπολογισμού του επομένου έτους που μοιάζει ότι θα είναι δύσκολο. Ο κύριος Σόμπες Μπέργκερ. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά. Κυρία Πρόεδρε, ανακεφαλαιώσατε εξαιρετικά όλες τις τροπολογίες. Δύο θέματα για την 10. Θα ήταν ίσως χρήσιμο να υπάρχουν κονδύλια πιστώσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και κυρίως βέβαια αυτό το θέμα του διπλασιασμού δεν είναι ρεαλιστικό. Είναι δύσκολο να απορροφηθεί αυτό το ποσό. Ευχαριστώ. Αυτά τα δύο. Πολύ καλά, σας ευχαριστώ. Οπότε θα μπορέσουμε με βάση όλα αυτά να επανέλθουμε με λεπτομερέστερες προτάσεις και μια ενισχυ... μια ισχυρή, να δώσει μια ισχυρή γνωμοδότηση η Επιτροπή Απασχόλησης. Αύριο θα εγκριθεί η έκθεση. Εγώ αυτό που το οποίο θα κάνω τώρα, βλέποντας το σύνολο των τροπολογιών, κύριε Λιαρικ, δεν μου είπατε Δέχεστε να αποσύρετε την τροπολογία παρθμών 9. Θα μου το πείτε ίσως μέχρι αύριο. Τι λέτε. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Έχουμε ένα πρόβλημα όμως. Γιατί Δηλαδή υπά, ε, ε, αναπτύσσεται, εξελίσσεται η επισφάλεια στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να βρεθεί κάτι, να βρεθεί μια διατύπωση που να προσπαθεί να πει ότι αυτοί οι εργαζόμενοι που έχουν επισφαλίσει θέσεις εργασίας, προσωρινές ε, θέσεις, προσωρινές θέσεις εργασίας, θα έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα δεν είναι θέμα γνωμοδότησης για το θέμα αυτό. Να σας προτείνω το εξή. Επειδή θα ξανασχοληθούμε με την 21 της κυρίας Τούρουνεν, μήπως θα συμφωνούσατε στην νέα διατύπωση που θα προταθεί εκεί να εισαχθεί η έννοια της επισφαλής απασχόλησης. Μήπως μπορούμε να βρούμε έτσι μια διατύπωση σε αυτό το σημείο. Κυρία Τούρουνεν, θέλετε να κάνετε πρόταση εσείς ή να το αναλάβω εγώ. Θα το, θα το αναλάβετε εσείς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τη δική μου παρατήρηση και ε, τη δυνατότητα να λάβουμε υπόψη μας την αναφορά αυτή στην επισφαλή απασχόληση Αυτό είναι το πρώτο θέμα το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε. Κατόπιν, τροπολογία υπαριθμών 6. Υπάρχει προφορική τροπολογία, αντίθετη εξ όσων αντιλαμβανόμαστε. Θα ψηφιστεί. Τροπολογία 13 Και εδώ θα πρέπει η ομάδα να μας πει αν αποσύρει την τροπολογία θέλει να την ε, διατηρήσει. Οπότε βεβαίως θα καταψηφίσω διότι δεν θεωρώ ότι έχει νόημα επιπλέον στο κύριο Γιούβιν θα ε, προτείνω στην 18 να προσθέσει κάτι λαμβάνοντας υπόψη και τη 17 του κυρίου Όρη στην 21 τη δουλειά θα μου την κάνει η κυρία Τούρουνεν σημειώνω ότι συμφωνεί ο κύριος Τόμας Μάν για την 24 και τον ευχαριστώ θερμά και τέλος, για την 27, βλέπω την... Θα μπαίνει ο κύριος Φιλίπ Μπουλά και θα μπορέσει ίσως να διαυκρίνει μέσω προφορικής τροπολογίας το πεδίο της πρότασής του γιατί μου φαίνεται ασαφής. Αυτό που δεν αναφέρα και που πιστεύω ότι όλοι σκέφτεστε είναι ότι θα θέλαμε, θα ήθελα να προσεγγίσει η ομάδα Γκούε την κυρία Σαρτιέ για να και εγώ θα το κάνω βέβαια για να συντάξει μια προφορική τροπολογία στην 15 για το επίπεδο του Ταμείου ε, Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Οπότε, μετά από όλα αυτά θα ψηφίσουμε αύριο. Οπότε, φτάσαμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης κανονικά, όμως θέλω να σας, ε, να σας ανακοινώσω ότι ε, έχει, βρίσκεται αλλού η εισηγήτρια, οπότε περνάμε στην ενέα Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα, μια εμπορική ανισορροπία. Ο, ο συνάδελφος Dirk Στέρκ ε, δε, συμφώνησε να συζητηθεί ε, πριν από την προηγούμενη και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που κατάφεραν να υποβάλω τόσες πολλές τροπολογίες σε μία έκθεση μόνο πέντε παραγράφων. Άρα διαπιστώνουμε ότι τους ενδιαφέρει το εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Μπορώ να τις δεχτώ τις περισσότερες τροπολογίες. Η γνωμοδότησή μας δεν θα πρέπει βεβαίως να είναι τόσο ογκώδης ώστε να μην καταφέρνουμε να περάσουμε αυτό που θέλουμε να πούμε. Θα προσπαθήσω λοιπόν να συντάξω συμβιβαστικές τροπολογίες και στο άμεσο μέλλον θα έρθω σε επαφή με τους συναδέλφους για να δω αν μπορούν και εκείνοι να δεχτούν τις προτάσεις μου. Βεβαίως θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν σε μια τροπολογία υποθέσει κανείς ότι το άνοιγμα της ε, Αγορά της Κίνας στον καπιταλισμό είναι αυτό καθεαυτό κακό και έχει οδηγήσει σε οπισθοχώρηση της Κίνας δεν μπορώ να ε, συνδυαστεί αυτή η άποψη με τη βάση τη γνωμοδότησή μου. Αυτό συμβαίνει ε, με αυτούς που ε, διατυπώνουν θέση τελείως διαφορετική από αυτή που διατυπώνω εγώ στην έκθεσή μου. Άρα υπάρχουν κάποιες τροπολογίε που δεν θα μπορέσω σαφώς να συμπεριλάβω στη, στους συμβιβασμούς που θα προτείνω. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε ως Επιτροπή είναι να περιοριστούμε στα θέματά μας. Φυσικά υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που δεν θα μπορέσουν να ε, συμπεριληφθούν στην έκθεση. Δεν είμαστε φερρυπίν η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για τον σεβασμό των συνθήκων κοινωνικής πρόνοιας στη ζωή των ανθρώπων. Ε, υπάρχουν όμως άλλα θέματα που μπορούν να συμπεριληφθούν στην έκθεση, όπως αυτά που ανέφερε ο κύριος Τόμας Μαν. Το θέμα είναι επίσης της πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν είναι κάτι που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Ίσως λοιπόν η τροπολογία 25 που αναφέρεται στο σεβασμό των εξαγωγών. Εδώ μπορεί να πούμε κάτι για τον περιορισμό των εξαγωγών, αλλά και πάλι είναι δύσκολο. Δεν είναι θέμα της Επιτροπής Απασχόλησης να το πει αυτό, είναι θέμα της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Υπάρχουν και κάποιες ενδιαφέρουσες προσθήκες στην έκθεση που υπέβαλα, η τροπολογία του κ. Λάμπερτ ας πούμε Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό και σε ποιο σημείο θα συμπεριληφθούν όλα αυτά. Θα ενσωματωθούν δηλαδή. Πάντως τις επόμενες μέρες θα προτείνω συμβιβασμούς. Υπάρχει κάτι που με απασχολεί και πρέπει να μας πει η Κομισιόν την απόψή της. Όχι η Επιτροπή. Η Επιτροπή μας εδώ. Τι ζητάμε από την Επιτροπή. Αν ζητάμε την Κομισιόν κάποια πράγματα, ενώ ξέρουμε ότι δεν θα, δεν θα υπάρχει εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, δεν μπορούμε να πούμε ότι η Κομισιόν δεν μπορεί να συνάψει οποιαδήποτε συμφωνία χωρίς καταληκτικά ε, καταληκτικές ε, διατάξεις για κάποια θέματα της κινέζικης αγοράς είναι πράγματα που ξέρουμε ότι δεν θα γίνουν. Επίσης, η τροπολογία υπαριθμών 19 του κυρίου Γκαετάνου λάθος, του κυρίου Κοφεράτη λέει ο μιλητής. Αν ζητάτε να συμπεριλαμβάνουν όλες οι εμπορικές συμφωνίες δεσμευτικές ρήτρε που θα απαγορεύουν ρητά κάποια πράγματα, δεν μπορεί να στείλουμε την Κομισιόν με τέτοια εντολή να διαπραγματευτεί με τους Κινέζους. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Το θέμα είναι να πετύχουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Αυτή είναι η βάση της δουλειάς μας. Το να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ό,τι μπορούμε, τα, ό,τι περισσότερο μπορούμε, να βελτιώσουμε τη διαπραγματευτική μας θέση με τους Κινέζου και να βοηθήσουμε την Κίνα να προχωρήσει προς τα διεθνώς αποδεκτά κοινωνικά πρότυπα. Αυτά είχα να σας πω κυρία Πρόεδρε. Θα ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων και θα συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί τους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στην ε, μητρική μου γλώσσα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τον εισηγητή και περιμένω με ιδιαίτερη ανυπομονησία τις συναντήσεις που θα οργανώσουμε για να συντάξουμε την ε, γνωμοδότηση αυτή προς την Επιτροπή Ίντα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πολιτική μας γραμμή και συμφωνώ με τον εισηγητή όσον αφορά την, τον αριθμό των τροπολογιών που αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και υπάρχουν και κάποια πολύ ευαίσθητες, κάποιες πολύ ευαίσθητες τροπολογίες που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήθελα να σας πω ότι εγώ υπογράμμισα το θέμα της αλληλεγγύης αλλά και την προστασία των ε, εργαζομένων, των μεταναστών. Τόνισα τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, οι εταιρείες συγγνώμη, στην, ε, σε επενδύσει στην Κίνα, αλλά επίσης και για την ρήτρα της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Αυτά είναι θέματα τα οποία αφορούν την Επιτροπή Ίντα. Μιλάμε για μια γνωμοδότηση που έχει ένα πολύ ενδιαφέροντα χαρακτήρα, γιατί και ο τίτλος εδώ ε, αναφέρεται σε μια ερώτηση, ρητορική όχι δεν γνωρίζω βέβαια, αλλά νομίζω ότι ο μεγάλος αριθμός των τροπολογιών δείχνει το ενδιαφέρον που έχουμε για την Κίνα, που είναι ένας μεγάλος εμπορικός πρωταγωνιστής αν θέλετε στην παγκόσμια σκηνή. Η Επιτροπή, πιστεύω, η Κομισιό μάλλον, θα πρέπει να παίξει μαζί μας ένα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι θα πρέπει να ζητήσει την εισαγωγή μιας ρήτρα που να αφορά την κοινωνική διάσταση των συμφωνιών. Θα πρέπει να υπάρχει και μια κοινωνική ρήτρα δηλαδή με ιδιαίτερα ενδιαφέρον τις τελευταίες επαφές ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, ε, συγγνώμη, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας ε, και παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα συζητήθηκαν στον κοινωνικό τομέα. Πιστεύω ότι εδώ εγώ τονίζω ιδιαίτερα την μεγάλη έμφαση στον ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κοινωνικό τομέα όσον αφορά την, ε, τις σχέσεις μας με την Κίνα. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Προφανώς ε, θα μπορούμε να βελτιώσουμε αν θέλετε τις εμπορικές μας σχέσεις ε, και οι εμπορικές μας συμφωνίες με την Κίνα και θα βρούμε τον τρόπο για να εκφράσουμε σαφέστατα την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάνω στο θέμα. Ο κύριος Τόμας Μάν και η κυρία Λαουμπέρ μετά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Dirk Stacks σίγουρα μπορούμε ε, να πούμε πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε σε ένα σημείο όλα τα σημεία που μας ενδιαφέρουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για όλο τον κόσμο, ε, σαφώς. Έχω κάνει ε, μια τροπολογία για τα πνευματικά δικαιώματα, είναι η τροπολογία 25 νομίζω, ε, που θεωρώ σημαντικό. Αυτό που είναι επίση σημαντικό είναι αυτό το οποίο ελέγχθη τώρα, ότι θα πρέπει ε, να φροντίσουμε να μπουν οι κοινωνικές ρήτρες. Γιατί μας ενδιαφέρει η Κίνα, μας ενδιαφέρει γιατί είναι ένας μεγάλος ε, εμπλεκόμενος στην αγορά και όταν μιλάμε για εξαγωγές δεν μπορούμε να ε, το εξετάσουμε ανεξάρτητα από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχουν ε, οι κοινωνικές συνιστώσεις. η Κίνα είναι, ε, ε, μέλος, μέλος ε, του ΠΟΕ, για να είναι κανείς μέλος του ΠΟΕ θα πρέπει να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις. Και θα ήθελα επίσης μέσα στα πλαίσια ενός διαλόγου να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα και στην τροπολογία 27 ε, λέμε ότι θέλουμε να έχουμε ένα διάλογο που θα οδηγήσει σε αποτελέσματα, όχι που θα αποτελέσει ένα άλοθη ε, ώστε να υπάρξει μηδενικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση. Και στην τροπολογία 28 χρειάζεται ε, καλύτερη επίγνωση μεταξύ των πολιτών και θα πρέπει και οι ίδιοι ε, οι εργαζόμενοι ε, να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. είναι πολύ σημαντικός ο τομέας της πολιτικής της κοινωνικής διάστασης και είναι σημαντικός παράγον για το μέλλον. Υπάρχει ε, ε, και η δυνατότητα του να ε, προωθήσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και την επίγνωση των ίδιων των εργαζομένων ότι μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα κοινωνικά ζητήματα. Είμαι σίγουρος ότι μπορούν να προκύψουν σημαντικές ε, και χρήσιμες συμβαστικές λύσεις ε, που θα δίνουν την ε, σωστή άποψη της Επιτροπής Απασχόλησης. Είναι μια έκθεση που μπορεί να μπει σε καλό δρόμο και να μας δώσει ένα καλό αποτέλεσμα τελικά. Κυρία Λάμπερτ, ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη γνωμοδότηση και για τη βάση την οποία μας έχει προτείνει και για την προσέγγιση την οποία την ακολουθήσει. Βλέποντας τις τροπολογίες, όταν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ τροπολογιών, μπορεί να χάσουμε κάποια σημαντικά σημεία. Γι' αυτό θα είναι σημαντικό να έχουμε συμβιβαστικές τροπολογίες. Ε, τελικά, αυτό που θέλουμε να προκύψει είναι κάτι ξεκάθαρο που δεν θα χάνει όμως ε, ε, αυτά τα οποία υπήρχαν στις τροπολογίες. πολλά σημεία μπορούμε να επικρίνουμε σχετικά με αυτά που συμβαίνουν στην Κίνα για την αγορά εργασία, για τα, τη συνδικαλιστική της οργάνωση κλπ. Αυτό όμω που θέλουμε να επιτύχουμε είναι πώ μπορούμε να τα βελτιώσουμε αυτά. Και όπω έλεγε και ο Τόμα, θέλουμε να δούμε πώ μπορούμε κάποια θετικά σημεία να τα εντοπίσουμε και να τα ενισχύσουμε. Αυτό θα έχει κέρια σημασία. Διαφορετικά ένας διάλογος τον οποίο μόνο θα επικρίνουμε χωρίς να κάνουμε τίποτα επικοδομητικό δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Απλώς θα σταματήσουν να μας ακούν και εμεί το ίδιο θα κάναμε στη θέση τους. Και όταν εξετάσουμε τα διάφορα σημεία κριτικής που εκφέρουμε, άκουσα και μια συζήτηση για τον προϋπολογισμό, νομίζω πολλά από αυτά τα σημεία τα επικρίνουμε και στη δική μας πολιτική για την αγορά εργασίας. Μπορεί να υπάρχει διαφορά όσον αφορά την οξύτητα των προβλημάτων, αλλά ορισμένα σημεία τα ζητάμε και για μας. Ε, η κοινωνική ρήτρα τι ζητάμε, ε, πρέπει να ξέρουμε και τι ζητάμε ως ε, προδιαγραφές από την αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Η τροπολογία 4 νομίζω ότι ε, κάπως ταιριάζει με αυτά που είπαμε για την κοινωνική ρήτρα και με την τροπολογία 26 του Τόμας Μαν. Θέλουμε να υπάρχει ο μηχανισμός για να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Είναι σημαντικό το θέμα ε, των ε, της αλυσίδας εφοδιασμού και των υπεργολάβων γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία δίνονται σε υπεργολαβία επομένως αυτός ο μηχανισμός στην αλυσίδα εφοδιασμού μας ενδιαφέρει. Η κοινωνική ρήτρα είναι σημαντική όχι μόνο για τα όσα γίνονται στην Κίνα, αλλά και για τις επιπτώσεις που έχει η Κίνα σε άλλες χώρες, όπου έχουν ε, ε, έργα σε λειτουργία και στην Αφρική και σε άλλα μέρη της Ασίας. Είμαι σίγουρη λοιπόν ότι ε, θα υπάρξουν επικοδομητικές συμβιβαστικές τροπολογίε. Θα ήθελα κι εγώ να συμμετάσχω στην προσπάθεια διαμόρφωση κοινών λύσεων. κάποιες διαφορετικές απόψεις πάντα υπάρχουν. Δεν είναι καινούριο να το πω εγώ εδώ, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάτι που θα μας βρίσκει σύμφωνους. Να δούμε ποιες τροπολογίες ε, είναι προτιμότερες για αυτή τη γνωμοδότηση, που να είναι τροπολογίες ε, και να δούμε και ποιες τροπολογίες ε, θα ήταν καλύτερο να υποβληθούν στην Επιτροπή Εμπορίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Θα ήθελα να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις. Καταρχάς, θα ήθελα να ζητήσω από όσου υπέβαλαν τις διάφορες τροπολογίες και αναφέρομαι στον κύριο Τόμας Μαν και στον κύριο Κοφεράτη όταν αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, οι τροπολογίες αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ε, αλλάξουν τη διατύπωση του κειμένου που πρότειναν και ίσως θα έπρεπε να αναφερθούμε και στις αρμοδιότητες της Επιτροπής διότι προφανώς ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα εάν τα δούμε από την, υπό την ευρεία του έννοια αναφέρονται και για τα και στα κοινωνικά δικαιώματα και στα δικαιώματα εργασίας άρα είναι και θέματα της δικής μας Επιτροπής και μπορούμε να το δούμε λίγο. Επίσης, Δεύτερη παρατήρηση είναι μία συνέχεια αυτών που είπε και ο εισηγητής για την κοινωνική ρήτρα. Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που υπάρχει αυτή η εμπορική ανισορροπία, που είναι και ο τίτλος της νομοδότησης, αφορά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι ανταλλαγές με την Κίνα. Δηλαδή δεν υπάρχει αμοιβαιότητα και στα στοιχεία της αμοιβαιότητας είναι τα στοιχεία της αμοιβαιότητας που θα έπρεπε να, πάνω στα οποία θα έπρεπε να στηρίζεται η, η συναλλαγή. Γι' αυτό θα πρέπει να μιλάμε για δίκαιες ανταλλαγές και για ε, την έννοια της αμοιβαιότητας. Πρέπει να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση, διότι υπάρχουν και ευρωπαϊκές ε, εταιρείε ε, επιχειρήσεις ε, σήμερα που δυσκολεύονται πάρα πολύ να πουλήσουν, να πουλήσουν ε, τα προϊόντα τους στην Κίνα. Και δεν εντάχθηκε η Κίνα στον ΠΟΕ για αυτούς τους λόγους. Επομένως θα πρέπει αυτή η κοινωνική ρήτρα, η ειδική ρήτρα ε, να προσεχθεί ιδιαίτερα. Προφανώ ο εισηγητή είπε δεν πρόκειται η Κομισιόν να πάει να διαπραγματευτεί με την Κίνα για τι κοινωνικέ ρήτρε. Και ίσω να μην κατάλαβα καλά τι είπατε, αλλά πιστεύω παρόλα αυτά ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και εγώ θα πρότεινα να συμπεριλάβουμε ε, και τις ε, περιβαλλοντικές ρήτρε. Αλλά τέλος πάντων άλλοι συνάδελφοι θα ασχοληθούν με το θέμα. Ελπίζω θα το κάνουν τουλάχιστον. Επομένως, η πρώτη παρατήρηση είναι να ζητήσουμε από τους συναδέλφους να επαναδιατυπώσουν ε, την επαναδιαποτύπωσή τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικές και τα κοινωνικά δικαιώματα. Επίσης, για τα κοινωνικά δικαιώματα θα πρέπει να έχουμε την κατάλληλη διατύπωση και να καλέσουμε τους τον εισηγητή μέσω των συμβαστικών τροπολογιών να εισάγει την ιδέα, την έννοια της αμοιβαιότητας και των δίκαιων εμπορικών συναλλαγών γιατί αλλιώ θα ήθελα να κάνω ε, μια προφορική τροπολογία. Λοιπόν, δεν ζητάει Ευχαριστώ, κύριε τον λόγο. Ε, ε, θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή και ζητώ συγγνώμη αν δεν κατάλαβα καλά αυτά που είπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως. Υπάρχει κοινωνικός διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας Ε, και μάλιστα έντονες ε, ανταλλαγές, έντονες επαφές. Αλλά ως κοινοβούλιο, αν ζητήσουμε οι εμπορικές ε, συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας να περιλαμβάνουν δεσμευτικές ρήτρες προσεγγίζουμε το θέμα τελείως διαφορετικά από τη μορφή του κοινωνικού διαλόγου που αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με την Κίνα πραγματοποιούνται μια σειρά από εμπορικές συνομιλίες. Και όπως είπατε υπάρχουν θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικής ε, πρόνοιας κλπ. που είναι όλα σημαντικά. Το θέμα είναι λεπτό, προφανώς εμείς ως κοινοβούλιο τι μπορούμε να περιμένουμε από την Κομισιόν. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να υπάρχει διάλογος για κοινωνικά ζητήματα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Υπάρχει και αυτό είναι πολύ θετικό και μάλιστα πρέπει να ενισχυθεί ο διάλογος αυτός. Κάποιο το ανέφερε αυτό, δεν θυμάμαι ποιο, και το ζήτησε. Βεβαίω, από την πείρα μου η Κίνα ε, η Κίνα ε, κοιτάζει μας ε, όταν θέλει να οργανώσει θέματα κοινωνικής πρόνοιας κλπ. Υπάρχει μια σειρά από νομοθετικά κείμενα που αφορούν την εργασία που μοιάζουν, που έχουν συνταχθεί με πρότυπα πρότυπο την Ευρώπη. Κάποιοι Βρετανοί καθηγητέ τα έχουν συντάξει. Δεν θα πρέπει να αποφύγουμε τον κοινωνικό διάλογο με την Κίνα. Αντίθετα. Τώρα, για τι υπόλοιπε τροπολογίες επιμένουν οι συνάδελφοι ότι οι ευρωπαϊκές επιχείρησεις πρέπει να τηρούν τους κανόνες στις συναλλαγές με την Κίνα. Το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή δεν είναι με τις ξένες επιχειρήσεις που επενδύουν στην Κίνα αλλά με τις κινέζικες επιχειρήσεις ή ίσως τις ε, ταϊβανέζικες και λοιπά επιχειρήσεις που επενδύουν στην Κίνα. Αν εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ε, θα πάνε όλα καλά στην Κίνα αν οι δικές μας επιχειρήσεις ε, ε, απλώς τηρούν τους κανόνες, κάνουμε λάθος. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους επί που θα υποβληθούν τις επόμενες ημέρες. Θα προσπαθήσω να δουλέψω αυτούς τους συμβιβασμούς, να συμπεριλάβω όσο το δυνατόν περισσότερο τις ιδέες σας Ίσως ε, οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου δεν θα μελετήσουν τόσο καλά την ε, γνωμοδότησή μας εάν συμπεριλάβουμε κάποια από αυτά τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ όλους. Ε, ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Ίσως θα έπρεπε να είχα πει και την αρχική μου ε, ομιλίας. Σας ζητώ να μελετήσετε τις 33 ε, και 56 του κυρίου Έλμερ που μου φαίνονται αντιφατικές και ως εκ τούτου απαράδεκτες. Θα μου πείτε την άποψή σας όταν θα επανέλθουμε. στη συζήτηση για τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Κυρία Πρόεδρε, λέει ο Σέλμερ, αν μιλάτε για, α, για την ε, το αν και μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι τροπολογίες, αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι θέμα του Προεδρείου. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Εγώ βεβαίω μπορώ να βάλω την πρότασή μου στον κατάλογο ψηφοφοριών και από εκεί και πέρα αν εσείς πείτε ότι, δεν, ότι είναι απαράδεκτες οι τροπολογίες θα δεχτώ αυτό που μου λέτε. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο, στην, ακριβώς στην πρόθεσή μου αυτή. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε στις 15 Ιουνίου για το συμβιβασμό και στις 16 θα γίνει η ψηφοφορία. Η κυρία Γκέρλινγκ μπόρεσε να έρθει, την ευχαριστώ και της δίνω το λόγο για να μελετήσουμε τις τροπολογίες ε, στην έκθεση γνωμοδότησής της διαδικασίας αφαιρεγγιότητας στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιχειρήσεις. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τους σκιώδεις εισηγητές της έκθεσης αφού έγινε σχετικά ήσυχα η προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων δεν ανταλλάχθηκαν πολλές απόψεις δεχτήκαμε 15 τροπολογίες για μια πολύ σύντομη γνωμοδότηση. Οπότε αποδεικνύεται ότι ε, το έργο αυτό είναι κάπως δυσκολότερο από ό,τι αρχικά είχα σκεφτεί, είχα υπολογίσει. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι με τη βοήθεια και των σκιωδών καταφέραμε να καταλήξουμε σε κάποιες λογικές και σωστές ε, συμβαστικές λύσεις παρά το ότι στην αρχή είχα θεωρήσει ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να συμβιβαστούν. Υπάρχουν όμως και κάποια θέματα. Η έκθεση έχει κάποια σύνθετα ζητήματα και έγιναν κάποιες συζητήσεις που νομίζω αξίζει τον κόπο να σας μεταφέρω. Πρώτον, δεν υπήρξε ακριβώς διαφωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει ζωντανή συζήτηση για το αν η δρομοδότηση αυτή εντάσσεται, είναι κατάλληλη σε σχέση με την κρίση, είναι σωστή σε σχέση με την κρίση, γιατί πολλά μέλη ε, επικεντρώθηκαν στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τη σχέση της με αυτήν ενώ άλλα μέλη θεώρησαν σαφώς ότι η έκθεση δεν έχει σχέση μόνο με την τρέχουσα οικονομική κρίση, αλλά ότι θα πρέπει να καλύπτει όλες τις δυνατές συνθήκες συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης και της ευημερίας που όλοι ελπίζουμε ότι θα εμφανιστεί στο μέλλον. Έγινε λοιπόν κάποια συζήτηση για το τι ακριβώς αφορά αυτή η γνωμοδότηση, αυτή η έκθεση και είναι λογικό πολλοί να σκέφτονται την κρίση, αλλά εμείς ελπίζουμε και προσπαθήσαμε να καλύπτεται και η ευρύτερη κατάσταση. Επίσης, συζητήσαμε σαφώς την, το δεύτερο συμβιβασμό που αναφέρεται διαμακρόν στο θέμα της αφαιρεγιότητας. από διάφορους χώρους υπήρξε η επιθυμία να διευκρινιστεί και να, καθοριστεί, να καθοριστούν οι όροι που αναφέρονται. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό μπορεί να γίνει εδώ. Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε με την ξεκάθαρη γνωμοδότηση και να μην εμπλακούμε ε, σε ένα τομέα που θα μας εμπλέξει και με τις αποφάσεις χιλιάδων ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Μάλλον με τις χιλιάδες αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Επίσης, θεωρώ ότι η διατύπωση στις συμβιβαστικές προτάσεις είναι θετική. Υπογραμμίσαμε ότι δεν θα πρέπει νόμος η νομοθεσία για την αφαιρεγγιότητα ε, να, να χρησιμοποιηθεί για να ε, μην ε, στην νομοθεσία, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη Δημιουργία Θέσεων Εργασία. Επίσης υπήρξαν συζητήσεις για την τροπολογία υπαριθμών 28. Εγώ ως εισηγήτρια, παρότι αυτό θα σήμαινε διαγραφή ενός μέρους τη έκθεσή μου, θα προτιμούσαν να υπάρχει υποστήριξη ε, στις τροπολογίες 25-27 και όχι μια ε, νέα τροπολογία 28. Όσοι συγγύτρια λοιπόν δεν έχω εμπλακεί σε αυτές τις συζητήσεις που από ό,τι καταλαβαίνω συνεχίζουν. Αυτά έχω να πω κυρία Πρόεδρε προς το παρόν. Σας ευχαριστώ κύριο Σαρκάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να σας εκφράσω τη συγγνώμη της σκιώσης ηγήτες της σοσιαλιστικής ομάδας η οποία βρίσκεται κάπου αλλού για σε μια ψηφοφορία αυτή τη στιγμή. Θέλω όμως εκ μέρους της να πω κάποια πράγματα. Καταρχήν, πρέπει να ευχαριστήσω την ε, κυρία Γκέρλινγκ, την Τζούλι Γκέρλινγκ, που επέδειξε πολύ ταλέντο σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις που έγιναν κυρίως όσον αφορά την τροπολογία Β. Πραγματικά ε, χρειάστηκε να διακηρύξει παντού και σε όλους ότι δεν μπορεί να, υπάρξει κοινός, να υπάρχουν κοινείς κανόνες για την απασχόληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μα δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε σε κοινωτικό επίπεδο όταν προσπαθούμε να, αντί να προχωρήσουμε διακυβερνητικά, να τους βάλουμε όλους στον ίδιο δρόμο. Ε, Συλλογικέ διαπραγματεύσει, συνταξιοδοτήσει κλπ. Δεν θα πρέπει να, θα πρέπει να διαγράψουμε αυτή την τόσο κατηγορηματική αναφορά. Και ίσως αργότερα να ασχοληθούμε με τον τόσο ακανθώδη αυτό κανόνα για την ευθυγράμμιση των επαγγελματικών θεμάτων στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό, διότι αλλιώς να επιμείνει η συγκίτρια σε αυτό, γιατί η ομάδα μας θα δυσκολευτεί να συμφωνήσει. Επίσης, όσον αφορά τον συμβιβασμό σε γάμα, ε, έχουμε πρόβλημα, κυρίως ε, με την τελευταία φράση. Υπάρχει μια διατύπωση ιδεολογική που δεν θα μας οδηγήσει πιθανά. Δεν θα ψηφίσουμε την τελευταία φράση. Τώρα, η συζήτηση ήταν πολύ επίκαιρη και ε, θα θέλαμε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε χωρίς καμία επιφύλαξη αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γέρλιν για την ε, έκθεσή της αλλά και για τις τροπολογίες με τις οποίες είμαστε σύμφωνοι σε γενικές γραμμές και να τη συγχαρούμε και για την πρόοδο που επετέφθη όσον αφορά την αρχική θέση της. Δηλαδή η συμφώνησε μαζί μας ότι η οδηγία αυτή βοηθάει ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα αφαιρεγγιότητας και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ε, τον καιρό της κρίσης, όμως η οδηγία αυτή πρέπει να ξεπερνάει την περίοδο της κρίσης και πιστεύουμε ότι μια βελτίωση της οδηγίας είναι εφικτή χωρίς όμως να αγγίξουμε τα κεκτημένα. Αυτό ήταν το πρώτο μας ε, σημείο διαφωνίας αν θέλετε γιατί εμείς θέλαμε να, υπάρχει μια, να υπάρχουν προτάσεις εναρμόνισης της νομοθεσίας, διότι αν θέλουμε να αναφερθούμε στην αφαιρεγγιότητα και να την ε, εξαφανίσουμε, θα πρέπει να Θα πρέπει να υπάρχει μια εναρμόνιση της ομοθεσίας η οποία είναι το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να εξασφαλίσουμε. Ε, η εισηγήτρια ήθελε να υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να γίνει μια απόπειρα εναρμόνισης. Εμείς όμως ε, θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε μια νομοθεσία που να στηρίζεται, που να βασίζεται στην εναρμόνιση. Ε, αυτό, ο στόχος μας ποιος είναι να προστατεύσουμε τον ε, αμοιβόμενο εργαζόμενο. Τον εργαζόμενο ο οποίος εισπράττει τον μισθό του. Τους μισθωτούς δηλαδή. Προφανώς ε, υπάρχουν και κάποιες, ε, κάποιες νομοθεσίες στα κράτη-μέλη τις οποίες δεν μπορούσαμε να αγγίξουμε. Π.χ. το δίκαιο της εργασίας. Όμως ζητάμε να σκεφτούμε λίγο παραπάνω τα θέματα εναρμόνισης έτσι ώστε να εξετάσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες κάποιες διαδικασίες, παραδείγματο χάρη το είδος και το ε, ύψος των αποζημιώσεων, το επίπεδο των εγγύσεων, οι προθεσμίες ε, που προβλέπονται από την διαδικασία και ο συντονισμός, η κεντρική ρύθμιση αν θέλετε των διαδικασιών έτσι ώστε να μπορούμε διασυνοριακά να ενημερώνουμε για τις διαδικασίες εφαρεγγιότητας. Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες για τις τροπολογίες που έχουμε υποβάλει και συμφωνούμε με την κυρία Γκέρλινγκ ε, με κάποιες από τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι οι λόγοι που μας ανάγκασαν να υποβάλουμε τις τροπολογίες μας και θα υποβάλουμε και κάποιες άλλες ακόμα. Γιατί θέλουμε να βελτιωθεί κάπως περισσότερο η όλη διαδικασία για την αφαιρεγγιότητα. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Περές. Ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Ο κύριος Κασί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ την κυρία Γκέρλινγκ για την έκθεσή της. Οι διαδικασίες αφαιρεγγιότητας είναι ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολιτικά εκρηκτικό μερικές φορές κατά τη διαδικασία της κρίσεως. Πολλά κράτη-μέλη έχουν αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα και εμεί ω πολιτικοί καταλαβαίνουμε τα προβλήματα των εργαζομένων που έχουν χάσει τη δουλειά του και που ε, μένουν χωρί εισόδημα επί μήνε πολλέ φορέ. Πρέπει να έχουμε όμω κατά ότι δίνουμε μια γνωμοδότηση για ένα νομοθετικό κείμενο που θα έχει επιπτώσει και μετά την κρίση, όχι μόνο κατά τη διάρκεια τη κρίση. Οι διαδικασίε αφαιρεγκαιότητα ε, μπορεί αυτέ καθ' να μην είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εκεί όπου που μπορούμε και εκεί όπου υπάρχει πολιτική βούληση θα κάνουμε αυτό το οποίο θεωρούμε καλύτερο για την ε, κοινή μας αγορά και για τους ε, εργαζομένους. Σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Όταν χρεοκοπεί μια εταιρεία, οι πιστωτές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι μέτοχοι όλοι αυτοί που έχουν επενδύσει πόρους με την πρόθεση να αποκομίσουν κάποιο κέρδος ε, για τον κίνδυνο στον οποίο ε, ε, εισήλθαν έχουν απώλειες. Όταν οι εργαζόμενοι πάνε στη δουλειά τους επενδύουν χρόνο και εργασία. Όλοι λοιπόν πλήττονται. Με τις τροπολογίες μας προσπαθούμε να έχουμε κάποιο συντονισμό που δεν υπάρχει δυνατότητα εναρμόνισης των διαδικασιών για να έχουμε ίση μεταχείριση των πιστωτών και μεταξύ αυτών ε, η συμμεταχείριση και για τους εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ζητάμε να δοθεί προτεραιότητα στους εργαζομένους στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Δεν βλέπω να θέλει κανείς το λόγο και δίνω ξανά το λόγο στη συνάδελφο την κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ. Θα συζητήσουμε με την ε, κυρία Χένια για το θέμα που αναφέρθηκε στην αρχή, γιατί κάπως πολύπλοκο μου φαν, κάπως μπερδεύτηκα. Θα προσπαθήσω εκτός συνεδρίασης να το συζητήσω μαζί της. Ε, για την τροπολογία 28 ε, θα ήθελα ε, να αναφέρω σε σχέση και με αυτό που είπε ο κύριος Μπουλόν ότι ε, η τροπολογία του είναι πολύ λεπτομερής. Συμπεριλαμβάνει τα μπόνους, τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τις παροχές. Δεν ξέρω αν είχε την πρόθεση να είναι πλήρης, πάντως είναι λεπτομερέστατη αυτή η τροπολογία. Η δική μου προσέγγιση είναι διαφορετική, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι εδώ ο κατάλληλο χώρο για να είμαστε ρυθμιστικοί σε τόσο λεπτομερέ επίπεδο. Όπω είπα όμω ήδη, συμφωνώ ότι όταν οι εργαζόμενοι βρίσκονται στην ατυχή θέση του να δουλεύουν για μια εταιρεία ε, η οποία καθίσταται αφαιρέγγια, θα πρέπει να έχουν αυξημένη προτεραιότητα. Δεν είναι θέμα προστασίας της απασχόλησης. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να συστήσουμε στην Επιτροπή Τζούρι να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στους εργαζομένους μέσα στον κατάλογο των πιστωτών. Και αυτή η προσέγγιση νομίζω ότι είναι κάπως διαφορετική. θα προτιμούσα τη δική μου τροπολογία 50 που λέει ποια είναι ξεκάθαρα ποια είναι ξεκάθαρη η δική μας προτίμηση, ότι θέλουμε δηλαδή η Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη σημασία στους εργαζομένους στο πλαίσιο όλων των πιστωτών αυτό το επίπεδο εναρμόνισης θα ήταν το ευκταίο και θα ήθελα η Επιτροπή μας προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθεί της δικής μου τροπολογίας 50 δηλαδή και όχι στο πλαίσιο της τροπολογίας ε, του κ. Μπουλόν που είναι λεπτομερέστατη γιατί όταν ε, δίνουμε ένα κατάλογο περιπτώσεων ε, είναι πολύ δύσκολο να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε καλύψει όλα. Πάντως, στα περισσότερα από αυτά τα σημεία, νομίζω ότι κινούμεθα προς πολύ λογικές συμβιβαστικέ λύσεις και θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας μέσα στις επόμενες ημέρες. Ε, très bien. Donc, je comprends que vous allez vous rapprocher de Madame Régnier pour vérifier comment est-ce que sur les amendements de compromis on peut euh, encore améliorer la, la situation. Et... Euh, Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ξέρουμε ότι θα κάνετε κάθε προσπάθεια για να βελτιώσετε το κείμενο και αύριο θα ψηφίσουμε τις 10 συμβαστικές τροπολογίες. Όπως σας είχα πει στην αρχή της συνεδρίασης, τώρα θα περάσουμε στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης. Και εδώ θα ήθελα να σας παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης που πρέπει να στείλει η Επιτροπή μας στην Επιτροπή Ήτρα ε, για το θέμα της ασφάλειας ε, των ε, υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Οκτώβριο του 2010 που ακολούθησε μετά ε, τον Απρίλιο του 2010 και το δράμα το οποίο διαδραματίστηκε στον κόλπο του Μεξικού ε, όταν ε, είχαμε έκρηξη στην εξέδρα γεώτρησης ε, σε κοιτάσματα πετρελαίου Deepwater Horizon. δεν εκφράστηκε άποψη κατά των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, ε, ε, αλλά εξάγουμε τα συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας, ούτως ώστε να έχουμε το απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας. Πολύ συχνά τα ατυχήματα αυτά συνδέονται με κάποια ανθρώπινα σφάλματα. Δεν μπορούμε να δαμάσουμε τη φύση, αλλά πολύ συχνά ανθρώπινες αποφάσεις βρίσκονται πίσω από τέτοια ατυχήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση γνωρίζουμε ότι δεν είχε σχέση με τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στην πλατφόρμα αυτή, όμως σίγουρα παίζει ρόλο η προσοχή που είχε δοθεί σε διάφορους δείκτες που είχαν υποτιμηθεί. Δεν ελήφθησαν υπόψη αποφάσεις, δεν ελήφθησαν αποφάσεις τη στιγμή που θα έπρεπε να ληφθούν γιατί εκτιμήθηκαν λάθος ορισμένοι δείκτες. Εδώ στις προτάσεις μας έχουμε 7 σημεία Ε, έχω ήδη λάβει σχόλια από τον οργανισμό του Bilbao που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και που υποστηρίζει βέβαια τη δική μας προσέγγιση με κάποιες συμπληρωματικές παρατηρήσεις τις οποίες θα σας αναφέρω. Η πρώτη παράγραφος της γνωμοδότησής μου αφορά τον ειδικό χαρακτήρα της εργασίας στις πλατφόρμες και τον κίνδυνο ανθρωπίνου σφάλματος προκύπτει ως εκ τούτου. Την προσέγγιση αυτή θα πρέπει να την συμπληρώσουμε μιλώντας και για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία και με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος της εφαρμογής. Και εδώ ακριβώς υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Και θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τη διαδικασία. Η δεύτερη παράγραφος της γνωμοδότησής μου μιλά για την οδηγία την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την πρόθεση να επανεξετάσει. Και εδώ ε, προτείνω τη μέγιστη και όχι την ελάχιστη εναρμόνιση. Σε ορισμένους τομείς μπορούμε να συζητήσουμε το είδος της εναρμόνισης που θέλουμε να έχουμε. Στο συγκεκριμένο όμως τομέα νομίζω ότι αξίζει τον κόπο ε, να ζητήσουμε τη μέγιστη εναρμόνιση. Στην τρίτη παράγραφο της γνωμοδότησής μου μιλώ για τους οργανισμούς επιθεώρησης Και στο σημείο αυτό επίσης ο οργανισμός του Μπιλμπάου θεωρεί ότι είναι χρήσιμο να υποβληθεί μια πρόταση. Στο τέταρτο σημείο της γνωμοδότησής μου αντικατοπτρίζεται το πνεύμα της Επιτροπής μας. Εάν θέλουμε καλή εφαρμογή των κανόνων υγείας και ασφάλειας, θα πρέπει να βασίζονται σε διαβουλεύσεις με τους εργαζομένους και σε συμμετοχή των εργαζομένων στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας. Η πέμπτη παράγραφος της γνωμοδότησής μου ζητάει από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να υπάρχουν απαιτήσει κατάρτισης για τους εργαζομένους με καθήκοντα υψηλού κινδύνου και ο οργανισμός του Bilbao έκανε την παρατήρηση ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή ε, ε, η προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. βέβαια το ότι πρέπει να υπάρχει μια τέτοια απέτηση σε παγκόσμιο επίπεδο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει εμείς να ξεκινήσουμε από τα του οίκου μας και να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε ευρωπαϊκές διατάξεις τις οποίες θα εφαρμόζουμε και θα εφαρμόζουμε και στα μη ευρωπαϊκά σκάφη που θα έρχονται σε ευρωπαϊκά ύδατα. Αυτό αξίζει τον κόπο να το τονίσουμε στο πλαίσιο της γνωμοδότησής μας. Στην έκτη παράγραφο προσπαθούμε ακριβώς για το λόγο που ανέφερα προηγουμένως ε, να τονίσουμε το ρόλο που παίζουν οι υπεργολάβοι. Το είδαμε όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο ατύχημα, αλλά και στην περίπτωση του Έρικα, Είδαμε ότι οι ελλείψεις προκύπτουν από την μη τήρηση κανόνων από τους υπεργολάβους. Σημαντικό λοιπόν το να ισχύσουν αυστηρά κριτήρια για τους υπεργολάβους. Και το τελευταίο σημείο είναι ένα σημείο στο οποίο ζητάμε οι εταιρείε με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζουν στις δραστηριότητές τους σε ολόκληρο τον κόσμο τους ίδιους κανόνες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων ένα θέμα που αφορά τη συμπεριφορά των πολιεθνικών και ένα σημείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Μια τελευταία παρατήρηση τώρα. Ο οργανισμός του Bilbao εφιστά την προσοχή μας στο ότι έχει ξεκινήσει μια έρευνα και δεν υπάρχουν ακόμη όλα τα συμπεράσματα από την έρευνα αυτή. Τα συμπεράσματα βεβαίω θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μα, αλλά αυτό δεν μα εμποδίζει να τονίσουμε τα σημεία που θεωρούμε σημαντικά. Αυτά λοιπόν ω παρουσίαση και θα δώσω το λόγο στον κύριο Τόμα Μαν καταρχήν και στην κυρία Λίν στη συνέχεια. Ο κύριο Τόμα Μαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση μου θυμίζει την συνεδρίαση στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο για τα 25 χρόνια από το Τσερνομπίλ και δεν ήταν θέμα μόνο της Επιτροπής Περιβάλλοντος ούτε ε, ε, άλλων επιτροπών και ε, εμάς ως Επιτροπή Απασχόλησης άμεσα μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα γιατί μας ενδιαφέρουν οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στους, αντιδρασ... στους πυρηνικούς αντιδραστήρες και μας ενδιαφέρει η κατάρτιση αυτών των ανθρώπων. Τι κατάρτιση έχουν πάρει, γνωρίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται και θα μπορούσε κανείς να πει ότι θεωρητικά είναι απλό. Έχουν κράνος, έχουν φόρμες ε, προστασίας, αλλά δεν είναι ε, αρκετό. Και όταν μιλάμε για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, χρειάζεται προηγούμενη κατάρτιση, χρειάζεται γνώση των κινδύνων τους οποίους διατρέχουν ε, και γνωρίζουμε ότι υπάρχει εκμετάλλευση πολλών εργαζομένων. Υπάρχουν πολλά ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση που φαίνεται ότι ο χρόνος εργασίας είναι απλώς θεωρητικός και υπήρχαν πάρα πολλέ καταγγελίες για τη μη τήρηση του ωραρίου εργασίας. Εμάς ως Επιτροπή Απασχόλησης πρέπει να μας απασχολήσουν αυτά τα θέματα. Είναι πολύ σημαντικό θέμα χρειάζεται χρόνος, ε, έλεγχος του χρόνου εργασίας ε, και κατάρτιση των εργαζομένων και θα πρέπει οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν ε, τους κινδύνους στους οποίους διατρέχουν και το πώς μπορούν να τους αποφύγουν. από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται εκεί ε, έχουμε ακούσει τα σχόλιά τους όταν είναι καλοκαίρι και ο καιρός είναι καλός ε, και ε, δεν υπάρχουν και μετεωρολογικοί κίνδυνοι είναι πολύ, πολύ διαφορετική η κατάσταση από ότι σε άλλες εποχές του χρόνου με πολύ πιο επικίνδυνες συνθήκες. Θα πρέπει να, εργάζ, να ελέγχονται επίσης, όπως είπε η κυρία Μπεχές, όχι μόνο ο, ο κύριος του έργου, αλλά και οι υπεργολάβοι. Θα πρέπει να ελέγχουμε τους υπεργολάβους που αναλαμβάνουν τμήματα του έργου και θα πρέπει όλοι να φέρουν την ευθύνη για το έργο το οποίο διεκπεραιώνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις σας και ελπίζω ότι και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Βιομηχανίας θα λάβουν υπόψη τα δικά μας μελήματα. Ευχαριστώ. Eh Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα που θέσαμε. Ιδίω λαμβάνοντας υπόψη όλες τις, ε, την, τον παγκόσμιο χαρακτήρα της επιχείρησης και γι' αυτό αυτό που προτείνεται η παγκόσμια πρωτοβουλία θα είναι πολύ χρήσιμο. Πρέπει να το επιδιώξουμε. Εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε από το ευρωπαϊκό. Ήδη υπάρχει κανονισμό για τους εργαζόμενους σε αυτές τις υπεράκτιες διαστηριότητες και, άλλες, και άλλα νομοθετικά κείμενα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να φροντίσουμε η ήδη φυστάμενη νομοθεσία να εφαρμόζεται σοβαρά και σωστά παντού. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εντοπίσουμε πού υπήρξε το ανθρώπινο λάθος γιατί θα γίνει σωστή η εφαρμογή της νομοθεσίας ένα μεγάλο μέρος της νομοθεσίας είναι πολύ αποσπασματικό και το παρακολουθούν διαφορετικές πλευρές. Πριν λοιπόν προχωρήσουμε με νέα νομοθεσία να δούμε την υφιστάμενη. Επίσης αναφέρεστε τη μέγιστη και όχι την ελάχιστη αρμόνιση. Ίσως αυτό να είναι πολύ περιγραφικό για την Κομισιόν η φυστάμενη οδηγία είναι αρκετά σύντομη και μιλάει για βασική υγεία και ασφάλεια. Δεν ξέρω αν πρέπει να προχωρήσουμε για την, ε, στην ελάχιστη εναρμόνιση, δεν το ξέρω. Αλλά το να επιβάλλουμε ε, ως Επιτροπή Απασχόλησης ε, κάποιους όρους δεν το θεωρώ σωστό. Επίσης μιλάτε για την ε, ε, για τους όρους εργασίας, τους το χρόνο εργασίας σε σχέση και με τις ε, επιχειρήσεις διάσωσης. Δεν ξέρουμε ε, αν γίνεται τώρα, τι ισχύει τώρα. Θα ήθελα να μάθω λίγο περισσότερα για το τι ακριβώς ισχύει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους ελέγχους που γίνονται από τα απαραίτητα από τα αρμόδια όργανα και αν δεν γίνονται, θα, έχετε δίκιο, θα πρέπει να δούμε. Αλλά πρέπει πραγματικά να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως τέσσερα, ναι στη συμμετοχή της, ε, των εργαζομένων. Απολύτως απαραίτητη. Αν δεν υπάρχει ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων, δεν θα υπάρχει τήρηση της νομοθεσίας. Απαιτήσει ε, εκπαίδευση ε, των εργαζομένων που εμπλέκονται σε αυτά τα, σε αυτά τα έργα βεβαίως και ε, αυτό το θέμα των υπεργολάβων είναι πολύ σημαντικό. Αν δει κανεί κάποια από τα ατυχήματα, μεγάλα ή μικρότερα, ε, οφείλονται στο ότι δεν έχουν ε, σωστά εκπαιδευτεί ή δεν έχουν σωστά τηρήσει οι υπεργολάβοι τους κανόνες. Επίσης είναι ενδιαφέρον να δούμε τη μελέτη του Μπιλμπάου. Περιμένω τα συμπεράσματά τους και τελικά η παγκόσμια πρωτοβουλία είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιδιώξουμε. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος που ζητάει το λόγο. Άρα να ευχαριστήσω τον κύριο Τόμας Μαν για την υποστήριξή του. Κυρία Ελίνε, για το θέμα μέγιστης εναρμόνισης. Ε, στο σημείο 1 υποστηρίζεται την ιδέα ότι το θέμα της εφαρμογής θα πρέπει να αναφερθεί. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ε, όντως, ένας από τους λόγους που η εφαρμογή δεν γίνεται με τον καλύτερο τρόπο είναι γιατί δεν ζητάμε την, μια μέγιστη εναρμόνιση. Ενισχύει μια μέγιστη εναρμόνιση εκεί όπου οι κανόνες είναι απόλυτα σαφείς. Εγώ πιστεύω ότι εδώ αυτή η μέγιστη εναρμόνιση μπορεί να είναι χρήσιμη. Τώρα για το σημείο 3 που αναφέρεται στους οργανισμούς επιθεώρησης να διαβάσω το σχόλιο της υπηρεσίας του οργανισμού του Μπιλμπάου τα θέματα ελέγχου και επιθεώρησης αποτελούν ένα ε, στοιχείο ενός ευρύτερου ε, πλαισίου που αφορά την, ε, τον όλο μηχανισμό ασφάλειας. Υπάρχει μια τέτοια απέτηση για όλες τις επιχειρήσεις και ακόμα και το να ζητάμε κάτι αντίστοιχο και για τις υπεράκτιες δραστηριότητες δεν είναι παράλογο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, για την συνεισφορά τους. Ε, ε, Επομένως, θα ήθελα να σας ζητήσω να υποβάλλετε όλες τις τροπολογίες σας, όχι πολλές, έναν λογικό αριθμό τροπολογιών. Είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε το σωστό αριθμό και μπορείτε να τις, να τις διατυπώσετε μόνο στα αγγλικά. Κάτι το οποίο θα περιορίσει και τον, ε, την ορμή, αν θέλετε, κάποιον να συντάξουν τροπολογίες. Λοιπόν, υπάρχει και η προθεσμία υποβολής ε, των τροπολογιών, 30 Μαΐου, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαδικασίες της Ήτρε. 5 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα. Επόμενη Δευτέρα, 5 η ώρα το απόγευμα. Και σας υπενθυμίσω ότι οι τροπολογίες αυτές ε, θα πρέπει να υποβληθούν στα αγγλικά. Και η, η Επιτροπή Ήτρε ψηφίσει στις 16, άρα θα πρέπει να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε στις 15 Ιουνίου. 15 Ιουνίου. Ωραία, ολοκληρώσαμε και με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, και απευθύνομαι στους συντονιστές. Αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσουν ε, μαζί μου ότι θα έπρεπε να διακόψουμε για ένα τέταρτο την συνεδρίαση και να ξεκινήσουμε την ε, ψήφιση της έκθεσης της κυρίας Λόπε Φοντανιέ, ούτως ή άλλως είναι και απούσα και καλό θα είναι να είμαστε συγκεκριμένοι την, όσον αφορά την ώρα που ξεκινάει η ψηφοφορία. Λοιπόν, και ζητώ συγγνώμη για τους παρόντες, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Ευχαριστώ.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 Λοιπόν, αν καθίσατε όλοι, έφτασε η 12 και μπορούμε να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Επί του σχεδίου γνωμοδότησης της κυρίας Λοπέ Φοντανιέ για την συνοχή και τη στρατηγική για την πολίτη συνοχής μέχρι το 2013. Πέμπτη έκθεση Επιτροπής. Παράγραφος 1 έχουμε συμβιβασμός α που υποβάλλουν πολλοί συνάδελφοι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατόπιν τροπολογία 13 Τόμας Mann κατά Λοιπόν, τροπολογία 13, μετά την παράγραφο 1, υπάρχει τροπο, προφορική τροπολογία της κυρίας Σρέτερ με σκοπό να ενταχθεί «Support the Commission in its aim to ensure and strengthening efficient and more visible ESF». Calls... mais ça peut être Δεν το βλέπω έτσι, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Ζητά από... Ζητά για το σκοπό αυτό η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν στο απαραίτητο ποσό ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στα διορθωτικά ταμεία. Εντάξει. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 14. Κυρία Τσίμερ και άλλοι. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 15 κυρίου Τόμας Μάνι. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, συμβιβασμός 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, κατόπιν τροπολογία 22 της κυρίας Φιγκερέντο υπέρ. Κατά αποχές θα επαλήθευση. Ε, δύο άτομα, εγώ και ο κύριος Φεγγανόφ δεν έχουμε την κάρτα μας. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Κύριε Κάμνοχ, είναι υπέρ και εγώ. Συν δύο δηλαδή. Ο κύριος Κάμνοχ και εγώ είμαστε υπέρ συν δύο. 24 υπέρ, 16 κατά εγκρίνεται. 23 του κύριου Τόμας Μαν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 Φιγκερέντο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 Τόμας Μάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 κυρία Φιγκερέντο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 Τόμας Μάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 Τόμας Μάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 Τόμας Μάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 ιδιοσυντάκτης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τρία, συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται φτάνουμε στην τροπολογία 33 της κυρίας Τσίμερ η οποία ε, συντάσσεται με το συμβασμό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται κατόπιν παράγραφος 3 δεν, δεν είδα καλά λέτε. Δεν... Επαλήθευση λοιπόν. Βυσί θα ψηφίσετε όλοι πέρα ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 23 κατά, 3 αποχές. Πράγματι ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, 37 της κυρίας Φιγκερέντο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 3, 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 κύριε Κοφεράτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4 συμβασμός D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατόπιν το συμβασμό D44 της κυρίας Τσίμερ και λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4, μία 49 της κυρίας Σρέντλερ και, και άλλων σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπογραμμίζει έως best practice, τις βέλτιστες πρακτικές και χωρίς τη λέξη που υπάρχει στον κατάλογο ψηφοφοριών. Εν πάση περιπτώσει, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Φτάσαμε στην τροπολογία 50 του κ. Ταμασμάν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 Σρόντερ και άλλων, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 5, συμβιβασμός ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 Σρέτερ και άλλοι. Καταπίπτει. Όπως και η 59. Η 60 απεσύρθη, παράγραφος 5, τροπολογία 63, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 του κυρίου Τόμας Μάν υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση. Επαλήθευση για την 64. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. 29 υπέρ, 14 κατά, εγκρίνεται. 65 του ίδιου συντάκτη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 66 επίσης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 συμβασμός F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 της κυρίας Γκέρνς συμβιβάζεται με αυτή υπέρ αποχές κατά αποχές ή 75 μετά την παράγραφο 6 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 76 της κυρίας Σόντερ καταπίπτει, οπότε φτάνουν στο συμβασμό G, παράγραφος 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατόπιν, η συμβαστική τροπολογία H, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά, παράγραφος 7, η παράγραφος 83 τη κυρίας Φουντάνια, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 85 κυρία Φιγκερέντο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 86 τη κυρία Σρόντερ και άλλων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 87 ψηφίζουμε, ψηφίζουμε παλήθευση για αυτήν. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Λοιπόν, η 87 του κυρίου Κρίστενσεν υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός ΑΗ παράγραφος 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, 94 του κ. Κοφεράτη υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά την 8 τροπολογία 95 της κ. Γκόντς με αίτημα χωριστής ψηφοφορίας πρώτο σκέλος in accordance with the report. υπέρ αυτού του μέρους κατά αποχές εγκρίνεται και similarly to the compulsory use και gender equality υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 96 της κυρίας Ρέντερ και άλλων υπέρ κατά αποχές θα ε, παληθεύσουμε έναρξη ψηφοφορίας Πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 24 κατά, απορρίπτεται. Η 97 του κ. Τόμασμαν καταπίπτει. Ψηφίζουμε την 98 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 99, εγκρίνεται, εγκρίνεται λέει η πρόεδρος. 99 της κυρίας Σουρέντερ υπέρ, Κατά αποχέ εγκρίνεται. Ε, της ίδια συντάκτη 1 ε, ε, εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 3 των ιδίων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 4 των ιδίων συντακτών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 6 επίσης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 7 των ίδιων συντακτών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 επίσης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για το σύνολο της γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 42 υπέρ. Με δύο αποχές συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και της δίνουμε την εντολή να μην ψηφίσει επί της ουσία η ε, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Λοιπόν, ραντεβού στις 3 κατά τα άλλα. Χαίρετε.